Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε πάλι. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Ντανιέλ Νουή, πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου που θεσπίστηκε στην ΕΚΤ στα πλαίσια του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού SSM. Σας είδαμε τελευταία φορά 19 Ιουνίου και η απόψινή συνάντηση είναι η τρίτη δημόσια κρόαση το 18. Και θα είναι η τελευταία τακτική ακρόαση με την κυρία Νουή υπό την ιδιότητά της ως ε, Προέδρου ε, του Εποπτικού Συμβουλίου. Θέλω να σας ε, ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για το εξαιρετικό έργο που επιτελέσατε όλα αυτά τα χρόνια στον εποπτικό μηχανισμό που ήταν μια δουλειά μεγάλη γεμάτη προκλήσεις η κοινή εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τεράστιο εγχείρημα και λίγοι προέβλεψαν ότι θα γινόταν τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά. Ένα τέτοιο ε, εγχείρημα δεν μπορεί να είναι τέλειο. Βεβαίως και υπήρχαν προβλήματα και εμείς ε, όπως είχαμε καθήκον ως κοινοβούλιο είχαμε πολλές ε, ζωντανές συζητήσεις για αυτά τα θέματα. Συνολικά όμως μπορούμε να μιλήσουμε για ένα επιτυχημένο εγχείρημα. Και μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλεται σε εσάς που προεδρεύσατε στο νέο αυτό θεσμικό όργανο και παρέσχετε αποτελεσματική εποπτεία των πιστοτικών ιδρυμάτων. Υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες εποπτείας, επιχειρηματικά μοντέλα και όλα αυτά έπρεπε να τα συγκεράσετε. Ακόμα πολλά μέλουν να γίνουν για να προχωρήσουμε προς μια ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση. Αυτό ε, απαιτεί ε, μεγαλύτερη εποπτική σύγκληση αλλά και νομοθετικό έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί για να έχει ο SSM τα εργαλεία που διαθέτει. Θα πρέπει να δούμε αν θα κινηθούμε και σε εθνικό επίπεδο προς την κατεύθυνση κανονισμού. Όλα αυτά είναι τα θέματα, τα θέματα μας. Ε, έχουμε και άλλα θέματα, τη Τραπεζική Ένωση, σίγουρα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ε, το ξέπλυμα χρήματος. Χαίρομαι γιατί πριν από τη συνάντηση αυτή, κατά το πρωί, κάναμε την συζήτηση για τον προληπτικό προστατευτικό μηχανισμό. Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε την νομοθετική διαδικασία μέχρι το τέλος του έτους ε, είναι μια ιδιαίτερα επιταχυμένη νομοθετική διαδικασία αυτή που ακολουθήσαμε για να συμπληρωθεί η λειτουργία του SSM και να μπορεί να δρά πολυπτικά και να παρέχει την απαραίτητη κάλυψη ε, ζημιών για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα με τον προστατευτικό μηχανισμό αλλά εμείς ε, στα πλαίσια της τραπεζικής δέσμης προσπαθούμε να οριστικοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερα θέματα. Ο τρίτος πυλώνας παραμένει ανοιχτός. Για το backstop, τον προληπτικό προστατευτικό μηχανισμό, ελπίζουμε να επιτελεστεί πρόοδος και είναι μια συνολική προσπάθεια που απαιτείται σε νομοθετικό επίπεδο, σε εποπτικό επίπεδο, σε τραπεζικό επίπεδο, αλλά αναγνωρίζω ότι ο SSM ήταν μια κινητήρια δύναμη για τη θέσπιση ε, μιας πιο ενοποιημένης τραπεζικής ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ και σας δίνω το λόγο για την παρουσίασή σας. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλου, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, Καθώ πρόκειται για την τελευταία μου ακρόση, όπω είπατε κύριε Πρόεδρε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την καλή συνεργασία στη διάρκεια ε, των τελευταίων πέντε ετών που σηματοδότησαν την θέσπιση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Θα εστιάσω σε τέσσερι τομεί βασικέ εξελίξει για τον κίνδυνο στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Χώρο για τις εποπτικές δραστηριότητες και για τα MPL, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και για τα ευρωπαϊκά τεστ αντοχής που προωθήθηκαν για την τραπεζική ε, ένωση αλλά και τη δράση για το ξέπλυμα χρήματος. Να ξεκινήσω με τον τραπεζικό τομέα στην Ευρωζώνη από την άποψη της εποπτείας. Ε, τα οι θεσμοί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησαν περαιτέρω την ανθεκτικότητά τους μέχρι το 2018. Οι τράπεζες που τις οποίες άμευσα υποπτεύει η ΕΚΤ διατηρούν μια ισχυρή κεφαλαιακή θέση με 14% περίπου ενώ χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν ε, ένα μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου τους για να ενισχύσουν τα ισοζύγια τους. Ε, συνεχίζουν να προοδεύουν ε, στη μείωση των αποθεματικών των μη εξυπηρετούμενων δανείων που είναι, ήταν και είναι προτεραιότητα για μας. Το 2018 η χονδρική αναλογία έπεσε στο 4% από το 7,5% στις αρχές του 2015. Παρά την στεναρή οικονομική ανάκαμψη και το τον όριμο επιχειρηματικό κύκλο στην Ευρωζώνη, τα σημαντικά θεσμικά όργανα παραμένουν στο 6,8% όσον αφορά τα χρεόγραφα κάτω από το 7,1% στις αρχές ε, τον προηγούμενο χρόνο. Οι τράπεζες της Ευρωζώνης είναι λιγότερο κερδοφόρες από ότι οι ομόλογές τους ε, στις ΕΠΑ λόγω ατελών προσαρμογών ε, στα επιχειρησιακά τους μοντέλα της και την υπερδυναμικότητα σε ορισμένους τραπεζικούς τομείς στην Ένωση. Ε, εάν δούμε το περιβάλλον, τον γεωπολιτικό κίνδυνο, ο οποίος έχει εντατικοποιηθεί ε, και ο πολιτικός κίνδυνος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί, έχουμε προβλήματα όσον αφορά την προστασία του εμπορίου σε κάποιες αναδυόμενες ε, Οικονομίες, νέα τιμολόγηση επίσης παγκόσμια επηρεάζουν αρνητικά τις δραστηριότητες στην Ευρωζώνη, άρα και τις τράπεζες. Επίσης η αύξηση ε, των ε, αποδόσεων των μονοετών ε, ομολόγων ήταν τελικά αρνητική εξέλιξη για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Ε, τώρα, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στον τομέα του πιστοτικού κινδύνου. Ιδιαίτερα διεξηγάγαμε μία ε, θεματική έκθεση για τις τράπεζες με το IVRS 9, ε, αυτό το πρότυπο, με στόχο οι τράπεζες να μειώσουν περισσότερο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε αυτό το επίπεδο έχει έχουν υποβληθεί στρατηγικές μείωσης των MPL στην ΕΚΤ, η οποία τα εκτίμησε ε, και με κοινέ εποπτικές ομάδες που έχουν ξεκινήσει εντατικού διαλόγους με τις τράπεζες για τις εφαρμογές αυτών των πλάνων για να προσφέρουν ενημερωμένη ε, κατεύθυνση, ενημερωμένα μάλλον κατευθύνσεις για την έξοδο από αυτό το πρόβλημα. Τώρα, για τη διαχείριση αυτού Έχουμε το τρίμα ε, όπως το ονομάζουμε ε, ε, εν συντομία. Έχουμε κάνει και τις σχετικές επισκέψεις. Περισσότερες από τις μισές τράπεζες που καλύπτονται από το ΤΡΙΜ έχουν λάβει τις πρώτες τους εποπτικές αποφάσεις. Συνεχίζουμε το διάλογο με τις τράπεζες σε σχέση με τον εμπορικό κίνδυνο για το επίπεδο 2 και επίπεδο 3 της έκθεσης και η ΕΚΤ έχει κάνει επισκέψεις σε επιλεγμένα σημαντικά ε, τραπεζικά ιδρύματα. Επίσης, ε, ε, συνεχίζουμε να εκτιμούμε το κίνδυνο κινδύνου μέσω του IT και να εκτιμούμε την ανθεκτικότητα των τραπεζών σε σχέση με σοκ ρευστότητας. Στις 2 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή δημοσίευσε τα πορίσματα ε, όσον αφορά τις δοκιμές αντοχής στις τράπεζες στο 70% των τραπεζών. 33 τράπεζες που άμεσα ελέγχθηκαν από την ΕΚΤ απεδείχθησαν πιο ανθεκτικές σε σοκ ε, τα τελευταία δύο χρόνια. Επίσης ε, κάναμε stress test στις τράπεζες που είναι άμεσα υπό εποπτεία και που δεν είναι κομμάτι του δείγματος της ε, Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, ε, μάλλον Τραπεζικής Αρχής, της ΕΜΠΑ. Ε, προσπαθούμε να εκτιμήσουμε και τις, ε, ε, τη ρευστότητα των τραπεζών όπως απαιτείται από τον κανονισμό εποπτείας. οι τράπεζες βασίζονται περισσότερο στα κεφάλαια από ό,τι πριν δύο χρόνια. Είναι στο 18,7% το 2018, ενώ ήταν στο 16,2% το 2016. Ε, επίσης, δυνατότητα απορρόφηση μακροοικονομικών σοκ αντικατοπτρίζεται στο τελικό αποτέλεσμα και εφαρμόζεται το πιο ε, σοβαρό δυνατό σοκ όπου έχουμε αύξηση εν μιας ποσοστίας μονάδας ε, από τα τελευταία δύο χρόνια. Εδώ έχουμε λοιπόν μια απόλυτα έτοιμη βάση που εξασφαλίζει πλήρως την εφαρμογή των ρυθμιστικών απαιτήσεων μέσα από τις μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι ενισχύ. Αυτό βέβαια θα πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και τα επίπεδα μη εξυπηρετωμένων δανείων που παραμένουν ανησυχία για πολλά ευρωπαϊκά ε, τραπεζικά ιδρύματα. Επιπλέον θα εξετάσουμε στενά τις προκλήσεις στη διάρκεια των φετινών stress test με ενόψη της βελτίωσης μελλοντικών ε, χρήσεων και θα κλείσω επαναλαμβάνοντας κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά για την εξασφάλιση μιας ομαλά λειτουργούσας τραπεζικής ένωσης και για την οποία εξαρτώμεθα από τη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου πριν και μετά τις ευρωεκλογέ. Έχουμε προχωρήσει πολύ χάρη στην ε, ε, τραπεζική εποπτεία όπω έχει δεσπιστεί, πρέπει ακόμα πολλά να γίνουν πριν ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση. Για το δέσμι για τι τράπεζε είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αναθεωρησία στη διάρκεια αυτή εδώ τη θητεία. Ξέρω ότι εργάζεται σκληρά επ' αυτού, κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλουμε ακόμα βελτιώσει κάποιου τομεί, όπω το το πιλωτικό ε, πλαίσιο 2 όπου θα εξετάσουμε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι τράπεζες, αλλά και τη δυνατότητα απορρόφησης αυτού. Επίσης, ε, όσον αφορά την μαζική εξάλληψη των MPL από τα αποθεματικά των τραπεζών, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό θα σταθεί στα πρότυπα που προτείνουν οι τράπεζες. Αυτή τη στιγμή αυτό καν δεν χρειάζεται, γιατί η σημερινή ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει κάποια ευελιξία όπου αυτό έχει νόημα. Ε, τέλος, θεωρούμε πως είναι σημαντικό να προβλέψουμε τις διατάξεις ε, ε, για οποιαδήποτε τράπεζα να ξεκινήσει η διαδικασία αφαιρεγγιότητας και εμπιστευόμαστε την έκτη για την εποπτεία των μεγάλων επιχειρήσεων και αυτό θα πρέπει να το δούμε μέσα στο πλαίσιο του Brexit. Τρίτον, όπως έχουμε ήδη ε, συζητήσει, χρειάζεται να έχουμε μία συγκεντρωμένη ε, ε, δράση για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος χρήματος υπό τη μορφή κανονισμού. Εργαζόμαστε επίσης για την εντατικοποίηση της προληπτικής εργασίας σε αυτό το τομέα, συντονίζοντας λειτουργίες μέσα στο πλαίσιο του SSM και το πλαίσιο της ε, εποπτείας ε, ε, και πάντοτε σύμμορφα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως ένας ενιαίος μηχανισμός όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις ΕΚΤ και τις αρχές καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος. Οι σχετικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται όσον αφορά τον εντοπισμό τραπεζών ε, των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο ευνοεί ξέπλυμα χρήματος. Επί τη βάση αυτή το Γραφείο για την Καταπολέμηση Ξεπλήματος Χρήματος θα ε, ασχολείται με τα συγκεκριμένα ε, και εντοπισμένα ζητήματα. Θα στρεωθεί επίσης ο δρόμος για τον καταμερισμό των δράσεων για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Χρειάζεται ρυθμιστική εναρμόνιση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε εθνικές ε, επιλογές, να βασιστούμε δηλαδή περισσότερο σε ε, κανονισμούς και οδηγίες που θα λειτουργήσουν ε, ομοιόμορφα και για τα θέματα ξεπλήματος χρήματος. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε δεχόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις και τώρα αρχίζουμε με τις ερωτήσεις και απαντήσεις ε, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, καταρχάς και θέλω να σας συγχαρώ για το τεράστιο έργο που ολοκληρώσατε ε, όντας επικεφαλής ε, του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας μπορέσατε να μετατρέψετε αυτό το νεοφιές ε, σχήμα σε έναν μηχανισμό που αναγνωρίζεται παντού στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Σήμερα διαπιστώνουμε στην Ευρώπη ότι το τραπεζικό σύστημα είναι ακόμα σχετικά κατακαιρματισμένο παρά όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και παρά τα επιτεύγματα όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση. Εξακολουθεί να υπάρχει λοιπόν μεγάλος καταμερισμός, κατακαιρματισμός και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πολλά, σε πολλά κράτη-μέλη ο τραπεζικό τομέα αποτελείται από μικρό, μικρά ιδρύματα τα οποία δεν είναι πάντοτε κερδοφόρα αποδοτικά, πράγμα το οποίο μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα προβληματικό. Για να ενισχυθεί, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας χρειάζεται να αναπτύξει πρωταθλητές που να είναι ευρωπαϊκοί πρωταθλητές και μέσα σε αυτήν την οπτική της ενίσχυσης της Τραπεζικής Ένωσης το ερώτημά μου είναι το εξής. Δεν θα ήταν επιθυμητό, ευκταίο να δούμε μια πιο δυναμική ε, παγίωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα ώστε να γίνει δε αυτή η παγίωση και η ολοκλήρωση δεν θα έπρεπε να προβλέψουμε κάποια στοιχεία του ευρωπαϊκού πλαισίου ε, όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας και τα καλά σας λόγια για το SSM. Όσοι έχουν ε, εργαστεί στα πλαίσια του SSM ε, χαίρονται πολύ όταν ακούνε τέτοια ε, θετικά σχόλια. Σε ό,τι αφορά τη τρέχουσα κατάσταση και την απαραίτητη ενίσχυση, πιστεύω πράγματι ότι πρέπει να εξελιχτούμε προς ένα ενιαίο μοντέλο προκειμένου να μας ε, βλέπουν ως ενιαίο τραπεζικό σύστημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε από πολύ διαφορετικά τραπεζικά συστήματα. Γιατί καθυστερεί τόσο η ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, η διάθεση των τραπεζών εκτεθούν σε κινδύνους, οι πιο ρηψοκίνδυνες ε, διασυνοριακές συναλλαγές δεν είναι τόσο ελκυστικές πλέον όσο πριν από την κρίση. Οι τράπεζες προσέχουν περισσότερο. Δεύτερον, δυστυχώς μετά την κρίση είδαμε κάποιες πρωτοβουλίες ring fencing και παραμένει ε, αυτό το καθεστώς και Αντιλαμβανόμαστε ακόμα περισσότερο χάρη στο SSM ότι η τραπεζική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει κατακαιρματισμένη. Υπάρχουν κανιά διαφορετικοί τρόποι ε, μεταφοράς των οδηγιών στο, ε, στα εθνικά δίκαια. Χρειαζόμαστε περισσότερες ε, ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι δυνατότητες διαφοροποίησης σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν στα πλαίσια μιας τραπεζικής ένωσης. Παρ' όλα αυτά, ισχύει όντω ότι χωρίς το τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, χωρίς το μηχανισμό εξασφάλισης των ε, το, χωρίς το μηχανισμό εγγύησης. Ε, αν σε εθνικό, ε, οι εθνικές ε, αρχές ε, θα αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις. Πρέπει να κινηθούμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως και εσείς πιστεύω πράγματι ότι χρειαζόμαστε μια ενίσχυση για πολύ απλό λόγο. Κάποιες από τις τράπεζες που ελέγχουμε δεν έχουν το απαραίτητο επίπεδο ιδίων ε, κεφαλαίων. Δεν είναι δικός μας ε, ρόλος να αποφασίσουμε ποιες συγχωνεύσεις πρέπει να γίνουν, ποιες προσεγγίσεις. Αυτό πρέπει να το αποφασίσουν οι τραπεζικές αρχές, οι επενδυτές, οι αγορές. Οι εποπτικές αρχές όμως παίζουν ένα πρωταρχικό ε, ρόλο. Καλούνται να ελέγξουν το νέο φορέα να εξετάσουν το επιχειρηματικό μοντέλο και να διασφαλίσουν ότι οι απαραίτητες συνέργειες ε, θα υπάρχουν, ότι ο νέος φορέας έχει ένα ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο κτλ και συνήθως αυτό είναι συνώνυμο προϋποθέσεων όρων που τίθονται προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των συγχωνεύσεων και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Οι ίδιες είναι οι προϋποθέσεις, είτε η συγχώνευση λαμβάνει χώρα σε εθνικό επίπεδο είτε διασυνοριακά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την παρουσία σας. Ε, εξ ονόματος των σοσιαλιστών θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για τη θέσπιση του SSM και τις προσπάθειες που καταβάλατε. Ε, ε, είπατε ότι ήταν μια εξαιρετική περιπέτεια, όπως και να είναι, ε, είστε ένας πυλώνας του τραπεζικού συστήματος. Έχουν, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα όμως. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό και μια και είναι η τελευταία φορά που συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Όταν ε, υποδεχτείτε τον, ε, το άτομο που θα σας διαδεχτεί τι ε, θα του πείτε, τι οδηγίες θα δώσετε ε, ανάλογα με την ε, εμπειρία σας και στα πλαίσια της συνεργασίας σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας. Κύριε Βουλευτή, πιστεύω σε ό,τι αφορά τη Τραπεζική Ένωση ότι πράγματι καταφέρουμε να μειώσουμε σημαντικά τους κινδύνους ε, για τις τράπεζες της Ευρωζώνης. Πολύ λίγοι λένε το αντίθετο. Ίσως κάποιοι πιστεύουν ότι δεν έχουμε επιτύχει αρκετά. Εγώ πιστεύω ότι ήχοι έχουμε κάνει πολλά. Υπάρχει μια όθηση, κυρίως σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Βλέπουμε κάθε μέρα ε, δημοσιεύσεις των ε, τραπεζών που προετοιμάζονται να ε, προχωρήσουν ε, περαιτέρω σε ό,τι ε, αφορά το ξεκαθάρισμα των ισολογισμών τους. Όπως και να είναι, δεν θα υπάρξει στιγμή όπου όλοι θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο κινδύνου, σε μηδενικό επίπεδο κινδύνου. Δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο, δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Πιστεύω επίσης ότι όλα αυτά είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης, γιατί αν συνέβαινε κάτι και αν ήταν απαραίτητη η ελληνική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε να μην βοηθήσουμε τη χώρα που, ε, την εκάστοτε χώρα που θα το χρειαζόταν, όπως ε, την περίπτωση της Ελλάδας για παράδειγμα. Η Ευρώπη ε, βοήθησε αυτό το συγγενή της που αντιμετώπιζε δυσκολίες. Και νομίζω ότι θα ήταν θετικό, υγιές, να ορίσουμε τις προϋποθέσεις της συνδρομής προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω η κίνδυνοι. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο τρίτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωση είναι απαραίτητος σε ό,τι αφορά το διάδοχό μου. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του. Εγώ έχω ακόμα έναν κατάλογο πραγμάτων που ε, παραμένουν και πρέπει να επιτευχθούν, ζητήματα που εκκρεμούν. Δεν θα μπορέσει να τα γνωρίσει αυτά τα ζητήματα ο διαδοχός μου. Σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση θα χρειαστεί να συνεχίσει τις προσπάθειες σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, προκειμένου να μην σταματήσουν απότομα οι θετικές ε, πρωτοβουλίες και σε ό,τι αφορά το TRIM θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Έχουμε ξεκινήσει ε, ε, κάποιες κινήσεις ε, προκειμένου να δούμε πώς θα χρειαστεί να εξελιχθεί η νέα νομοθεσία σχετικά με το ΣΡΕΠ. Και φυσικά θα χρειαστεί θα χρειαστούν και άλλε ε, προσπάθειες προκειμένου να προχωρήσει η Τραπεζική Ένωση σε ό,τι αφορά την εξυγίανση των ε, τραπεζών, γιατί και σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να είμαστε πιο Ευρωπαίοι. Ήμουνα πρόσφατα στο Βερολίνο και εξήγησα ότι μία ευρωπαϊκή απόφαση για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον να εξηγιανθεί μια τράπεζα αντί να διαλυθεί. Πρέπει πρώτα να απαντηθεί αυτό το ερώτημα και μετά να προχωρήσουμε παρατέρα. Αν υπάρχουν 19 τρόποι εξυγίανσης ε, λόγω των 19 ε, ε, τρόπων μεταφοράς του μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, τότε η απάντηση είναι όχι και οδηγούμαστε σε μια διάλυση. Και τότε αντιμετωπίζουμε πολλά και διαφορετικά ε, πλαίσια. Κάποιοι λένε ότι όχι, δεν θα ε, γίνει ε, διάλυση γιατί δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στη Λετωνία και στο Λουξεμβούργο έγινε αυτό. Γενικά, πάντως, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και η νομοθεσία. Ευχαριστούμε. Είναι πολύ καλή καλό αυτό το θεματολόγιο. Και για το τελευταίο προσπαθούμε να συμβάλλουμε και εμείς στην επίλυση, να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες που είχαμε. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο και αυτό, λέει ο πρόεδρος στην κυρία Μπερές. Αλλά και αυτό ήταν σημαντικό που προσπαθήσαμε να το λύσουμε και ήταν χρήσιμη και η συνεισφορά του SSM εδώ. Από ε, την ομάδα ECR δεν βλέπω. Ο Ραμόν Τρεμόζα για του Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Νουή, καλωσορίσατε ακόμη μια φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας εργασία όλα αυτά τα χρόνια. Θα μιλήσω στα αγγλικά για να θέσω την ερώτησή μου. Καταρχήν, να σας ρωτήσω κάτι για την, το άνοιγμα τραπεζών δημοσίου. Σε κάποια κράτη-μέλη η έκθεση στο δημόσιο των τραπεζών είναι πολύ μεγάλη, πέρα από την οικονομική, δημοσιονομική θέση της χώρας. Έτσι οι τράπεζες γίνονται ευάλωτες αν οι, ε, οι αγορές ε, θεωρήσουν ότι δεν είναι καλή οικονομική πολιτική. Μπορεί να υπάρξει νέα κρίση. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξουν ε, υψηλά όρια στα ανοίγματα. Και μια δεύτερη ερώτηση. Υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις σε ό,τι αφορά την ε, ε, καθάριση, την εξυγένση της μιας τράπεζας στη χώρα μου. πρέπει να ξαναδούμε τις λέξεις fail ή likely to fail, από την χάνει είναι πιθανόν. Αυτό εξετάστηκε και σε μια διάσκεψη 15 Οκτωβρίου. Οι ορισμοί αυτοί δημιουργούν πάρα πολύ δύσκολα ερωτήματα. Τι πιστεύετε για τους ορισμούς, πρέπει, δεν πρέπει να είναι πιο σαφείς. Ευχαριστώ πολύ. Για το δημόσιο κίνδυνο, το τωρινό ρυθμιστικό πλαίσιο αντιμετωπίζει το δημόσιο χρέος ως μηδενικού κινδύνου. Η ΕΚΤ παρακολουθεί το δημόσιο χρέος ε, ως μέρος της συνεχιζόμενης εποπτείας, αλλά η επανεμφάνιση ε, θεμάτων όπως βιωσιμότητα δημόσιου χρέους, ε, αυτό πράγματι μας απασχολεί. Πρέπει να πω ότι αυτό είχε συμπεριληφθεί στο τελευταίο stress test ήταν και στο stress test που έγινε το 2016. Οπότε προς το παρόν αυτό είναι ο πιο λειτουργικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Γενικότερα θα έλεγα ότι το ζήτημα είναι σημαντικό και πρέπει να εξεταστεί στον πυλώνα ένα καταρχήν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ΕΚΤ, έχει θέσει τέσσερις γενικές αρχές που πρέπει να έχουμε υπόψη ε, στη μεταρρύθμιση του πυλώνα 1. Οποιαδήποτε ρυθμιστική αλλαγή θα πρέπει να περάσει όχι από ποσοτικούς περιορισμούς αλλά από ε, επίπτωση στις τιμές. Θα πρέπει να προληφθούν σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά. Θα πρέπει το παγκόσμιο επίπεδο δεδομένου του ενδεχόμενου πρέπει να ληφθεί υπόψη το παγκόσμιο επίπεδο και οι ίσοι κανόνες του παιχνιδιού και θα πρέπει να υπάρχει μια μακρά μεταβατική περίοδος. Βέβαια, αν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση με τρόπο θετικό, αυτό είναι ένας τρόπος για να μειώσουμε την ε, διαπλοκή αυτή τραπεζών και δημοσίου. Σχετικά με τους ορισμούς, failing ή likely to fail, λέτε ότι ίσως οι ορισμοί πρέπει να επανεξεταστούν ή αναθεωρηθούν. Πιστεύω προσωπικά ότι ενιολογικά είναι καλή προσέγγιση και περιγράφεται καλά στην οδηγία. Ως επόπτες προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε μια ε, μεθοδολογία. Το failing είναι εύκολο, αλλά το likely to fail αυτό είναι η πιο σύνθετη ε, συνιστόσα του ορισμού. Προσπαθήσαμε να στηριχθούμε σε κριτήρια όμως για να δούμε τι είναι αυτό το likely to fail, τι σημαίνει για τη φερεγγιότητα, όχι τόσο για τη ρευστότητα, γιατί είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε μια κρίση ρευστότητας. Το, η φερεγγιότητα όμως και η αποτυχία, η πτώχευση λόγω φερεγγιότητας είναι πιο σύνθετο ένα θέμα. Γενικά είμαστε καλυμμένοι από τους ορισμούς γιατί πιστεύω ότι λειτουργήσαν καλά για τις τράπεζες που είπαμε ότι είναι failing ή likely to fail. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές δυνατότητες. Μπορεί να ε, καθαριστεί η τράπεζα ή μπορεί να εξηγιανθεί η τράπεζα αλλά αυτό είναι στα χέρια του ενιαίου ε, μηχανισμού εξυγένσης. Ο Σβέν Γκίγκολτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Νουή, πρώτα απ' όλα, εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων και ως ένας από τους δύο εισηγητές τότε που όλοι μαζί δημιουργήσαμε τον SSM θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη τη δουλειά που κάνατε. Αν αμφίβολα καταφέρατε να κατασκευάσετε έναν γνήσιο ευρωπαϊκό μηχανισμό και θεσμικό όργανο. Βέβαια, πολλές φορές οι διαφωνίες ε, είναι αναπόφευκτες, αλλά πάντοτε δράσατε με ακαιρεότητα υπέρ του ευρωπαϊκού συμφέροντος και πάντα δείξατε σεβασμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το είδα και σε δημόσιες ακροάσεις και κλεισμένων των θυρών και σας ευχαριστώ. Τώρα, ε, η συνήθιση δουλειά της ε, Επιτροπής μας είναι να κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις. Κυρία Νουή, ε, δεν πρέπει να φύγετε χωρίς δύσκολες ερωτήσεις. Πρώτον, όταν συζητάμε για το θέμα των ε, κόκκινων δανείων, πώς θα επιβάλλετε τους κανόνες σε μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εσείς ε, εξετάζετε πέρα από τις άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες και τις μικρότερες τράπεζες όπου υπάρχουν αμφιβολίες για το πώς ε, ε, εφαρμόζονται οι κανόνες. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Επίσης, το σκάνδαλο Cum-Ex από το κονσόρτσιουμ που αποκαλύφθηκε από τους δημοσιογράφους. Ε, δόθηκαν υποσχέσεις ότι στο μέλλον θα δρουν όλοι με αμεροληψία και ακαιρεότητα. Όμως συνεχίστηκε η κλοπή των χρημάτων των φορολογουμένων καταστρατηγώντας το φορολογικό δίκαιο και πολλοί βοήθησαν τον κόσμο να παραβιάσει τον νόμο. Το άρθρο 11 του κανονισμού του SSM σας επιτρέπει να διεξάγετε ευρωπαϊκές έρευνες. Δεσμεύεστε να, να προσπαθήσετε στο πλαίσιο της ε, λήψης αποφάσεων να δώσετε συνέχεια στο θέμα για να γίνει ευρωπαϊκή έρευνα ε, με, και να δείτε τη συμμετοχή των τραπεζών που εποπτεύεται στο σκάνδαλο αυτό Κουμέξ. Ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σας λόγια. Σχετικά με το παράρτημα αυτό για τα κόκκινα δάνεια έχετε δίκιο ότι παρόμοιους κινδύνους πρέπει να, να αντιμετωπίζουμε με παρόμοιο τρόπο στον ισολογισμό των τραπεζών και θα πρέπει να ε, ε, επιτυγχάνεται τέλος μια σύγκληση. Αυτό γίνεται και για τα παλαιά κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν δύο δυνατότητες ή να έχουμε μία ε, σταδιακή εφαρμογή του παραδείγματος στα θέματα των παλαιών δανείων και μετά βέβαια θα πρέπει να γίνονται αιτήματα κατά περίπτωση στην τράπεζα ή θα πρέπει να έχουμε περισσότερη εφαρμογή κατά περίπτωση των κανόνων. Δηλαδή με βάση την ικανότητα των τραπεζών να δημιουργήσουν κεφάλαιο και να προβούν σε πρόσθετες ε, προβλέψεις έχουμε ανάλογα κάποιες προσδοκίες τράπεζα Χωρίς να υπάρχει ένας γενικότερος στόχος phasing in. Αυτή είναι η λύση που προκρίθηκε οι τράπεζες λοιπόν εξετάστηκαν ως προς την ικανότητά τους να κάνουν αυτό το phasing in. Υπάρχουν διαφορετικές ομάδες τραπεζών, κάποιες ε, ε, ε, δουλεύουν πολύ πιο γρήγορα από άλλες και εξηγήσαμε στις τράπεζες τι περιμένουμε από αυτές. Και έτσι γίνεται η εφαρμογή τώρα και θα δούμε, θα έχουμε και άλλες προσδοκίες μετά από λίγα χρόνια, προχωρώντας κάθε χρόνο και βλέποντας ε, τι γίνεται. Αυτό το αντέντουμ λοιπόν, αυτό το παράρτημα ε, ε, θα πρέπει σταδιακά να εφαρμοστεί με phasing in σε θέματα παλαιών δανείων που θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τους ισολογισμούς των τραπεζών. Όχι για, Α, απάντησα για τα, τις σημαντικές. Για τη λιγότερο σημαντικές τράπεζες έχουμε επίσης ένα σχέδιο, αλλά θα εφαρμοστεί από τις εθνικές αρμόδιες αρχές με αναλογικότητα όπως όλα τα μέτρα που προέρχονται από μας. Με κάποια καθυστέρηση βέβαια σε σχέση με τις, τα σημαντικά ιδρύματα γιατί θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο κάποια από τα λιγότερο σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το αντέντουμ αυτό ισχύει και για τους δύο και για τις δύο κατηγορίες. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή πρέπει να το χρησιμοποιήσουν για τις ροές. Και το μετά θα ακολουθήσει το δεύτερο ή τρίτο βήμα, ανάλογα με το τι εννοούμε με τα βήματα, ε, θα πρέπει να γίνει και για το στόκ. Όλες οι αρχές, οι εθνικές αρμόδιες αρχές γνωρίζουν ότι το άντις ε, θα εφαρμοστεί, θα γίνει συνολικότερη εκτίμηση και λιγότερο αυστηρή για τις ε, ε, λιγότερο σημαντικές ε, τράπεζες αλλά θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσουν το αντέντουμ πρώτα για το, τη, στη, και μετά και στο ενεργητικό. Βέβαια, ε, το, το, το κούμεξ αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Ε, δεν ε, έχουμε τέτοιες αρμοδιότητες, δηλαδή δεν παρακολουθούμε τις καταστρατηγίες του ποινικού, της ποινικής νομοθεσίας. Πάντως, στηρίζομαι την κοινοβουλευτική έρευνα παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες που θα που χρειαστείτε. Και επίσης, αν έχουμε λόγους να υποπτώσουμε, πιστεύόμαστε ότι μπορεί να διεπράχθει ποινικό έγκλημα, τότε μπορεί να αναθέσουμε Τότε θα πρέπει να ζητήσουμε από την ε, οικία αρμόδια ε, εθνική αρχή να παραπέμψει το θέμα στο αναρμόδιο φορέα και να ε, ασκηθούν διώξεις ενδεχομένως βάσει του ποινικού δικαίου της χώρας δεν έχουμε αρμοδιότητα, αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές να δώσουν στον Εθνικό Εισαγγελέα ή στην ποινική δικαιοσύνη να δώσει τις πληροφορίες που χρειάζονται. Και εμείς παρέχουμε και προσφέρουμε τις πληροφορίες που έχουμε στη δικαιοσύνη ή στο κοινοβούλιο ανάλογα. Ευχαριστώ. Στις μικρές τράπεζες πάντως θα ισχύσει το ε, addendum του πυλώνα 1 και θα ισχύσει ο προστατευτικός μηχανισμός. Θα έχουμε δηλαδή τα, πρόσθετα μέτρα του πυλώνα 1. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Νουή, θα ήθελα και εγώ εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας, αλλά και εκ μου προσωπικά, να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε, καθώς είναι η τελευταία σας παρουσία με την σημερινή σας ιδιότητα στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Το πρώτο, σημειώσατε ότι έχει γίνει στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων και της θητείας σας μια μεγάλη μείωση των κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα. Θα συμφωνήσετε όμως μαζί μου ότι δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό βήμα για την παράλληλη αμοιβεοποίηση των κινδύνων. Γιατί το ίντις, η πρόταση της Κομισιόν, που υποστηρίζεται από, μια, ε, από ένα πολύ ευρύ φάσμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, επειδή είπατε ότι υποστηρίζετε την άποψη ε, ότι πρέπει να προχωρήσει το ίντις, τι συμβουλή θα δίνατε επ' αυτού στον διάδοχό σας τον κύριο Ενρία. Η δεύτερη ερώτηση, παρότι σημείωσα την απάντησή σας στον συνάδελφο Γκίγκολτ ότι δεν ασχολείστε με τις ποινικέ υποθέσεις, το πρόβλημα παραμένει το μεγάλο σκάνδαλο Κάμεξ, μέσω του οποίου εκλάπησαν από τα δημόσια ταμεία και από τις τσέπες των συνεπών φορολογουμένων δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, πέρασε κάτω από το ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών. Το βρήκαν μερικές δεκάδες δημοσιογράφοι και απέτυχαν να το βρουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Επομένως, πώς θα καλυφθεί αυτή η μαύρη τρύπα. Δεν αρκεί να δίνετε πληροφορίες στις κοινοβουλευτικές επιτροπές που τη ζητούν. Το θέμα είναι πώς θα κλείσουμε την τρύπα μέσα την οποία περνούν τέτοια σκάνδαλα τα οποία ανακαλύπτουν στη συνέχεια κάποιοι whistleblowers και όχι οι φύλακες των θεσμών που είσαστε εσείς. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι υπάρχουν κάποιες προτάσεις για την διαχείριση και την μείωση των κόκκινων δανείων στην πατρίδα μου την Ελλάδα που έχουν διατυπωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα ήθελα να μου πείτε αν, έχετε, αν τις έχετε δει και αν έχετε κάποιο σχόλιο από αυτόν. Ευχαριστώ. Regarding EDIS Για την αμοιβιοποίηση του χρέους σε κάθε συνάντηση που πηγαίνω λέμε ότι το ΕΝΤΙΣ πρέπει να ε, τεθεί σε ισχύ για μειωμένο, και έχουμε, μειωμένο, έχουμε μειώσει τον κίνδυνο αρκετά για να προχωρήσουμε. Θα έχουμε πρόοδο στο ΕΝΤΙΣ και ο διαδοχός μου θα πει το ίδιο. Αυτό είναι ο ρόλος της ε, ΕΚΤΕ. αλλά η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί πρώτα σε πολιτικό επίπεδο. Ε, δεν μπορούμε εμείς να δράσουμε αυτόνομα. Αλλά σίγουρα ε, έχετε τη μεγάλη υποστήριξή μου για αυτό το project. Θα ωφελήσει όλους γιατί εμείς δεν επιλέγουμε να μην αναλάβουμε το κόστος, οπότε πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός. Τώρα, για το ποινικό θέμα του Κάμεξ και παρόμοια δικήματα, Αυτό είναι πολύ τεχνική δουλειά γιατί χρειάζεται φορολογικός έλεγχος και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πολλούς ειδικού ε, για τα φορολογικά καθεστώτα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα από τους φορολογικούς ελεγκτές για να ανακαλύπτουμε τέτοια προβλήματα. Σε μία επιθεώρηση επιτόπου όμως, όταν για παράδειγμα υποπτευθούμε ότι κάτι τρέχει που μπορεί να είναι ποινικό αδίκημα, εκεί πράγματι φροντίζομαι οι πληροφορίες να παρέχονται στις ε, φορολογικές αρχές, στις αρχές ε, καταπολέμησης του ξεπλήματος ε, και παλιά είχε συμβεί να ανακαλύψουμε πριν από τους εφοριακούς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ότι υπήρχαν κάποιοι μηχανισμοί που παρακάμπτονταν. Αλλά γι' αυτό το σκάνδαλο Κάμεξ πράγματι ε, δεν το προλάβαμε το πρόβλημα. Το είδαμε αφού είχε ε, εκδηλωθεί και οι πληροφορίες δόθηκαν ε, στις εθνικές αρχές. Και όταν μας ζητήθηκε δώσαμε πληροφορίες για το κοινοβουλευτική έρευνα. Α, και τα κόκκινα δάνεια. Ξέρω ότι κάτι γίνεται. Όταν συζήτησα με τους συναδέλφους της Τράπεζα της Ελλάδας, μου είπαν ότι ακόμα συνεχίζεται, συνεχίζονται οι εργασίες και δεν έπρεπε να γίνουν διαρροές, δεν έπρεπε να διαρρεύσουν τόσο γρήγορα. Δεν υπήρχε χρόνος για να μας ενημερώσουν καλύτερα. Μπορεί να είναι ένα σύστημα όπου οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα το δικό τους κομμάτι των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να τα ε, υποβάλουν στην εταιρεία διαχείρισης των ε, περιουσιακών στοιχείων που θα χρηματοδοτείται μέσω φορολόγησης. Και η τράπεζα θα κάλυπτε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και τα ε, χρήματα για την κάλυψη μεγαλύτερων συναλλαγών. Δεν ξέρω όμως περισσότερα, είναι σύνθετο το θέμα είναι δημόσιο χρήμα, μπορεί να είναι δημόσιο χρήμα που βρίσκεται στην τράπεζα, οπότε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα πρέπει να το δει το θέμα. Πάντως είμαστε ακόμα στην αρχή. Είναι εργασίες εν εξελίξη. Δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο. Έχω απλώ τηλεφωνικές επαφέ με τους συναδέλφους μετά από τις ειδήσει που διάβασα στις εφημερίδες και τους ρώτησα. Δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση να σας δώσω. Σίγουρα όμως τις επόμενες εβδομάδε θα μάθουμε περισσότερα. Ευχαριστώ κύριο Κίρσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Νουή για τις προσπάθειές της και την συμβολή της Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα. Νομίζω ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ Ρώμης και Βρυξελών και αυτός ο ανταγωνισμός θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές. Αυτή είναι η στρατηγική της Ιταλικής κυβέρνησης από ό,τι καταλάβαμε και φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες αντιδρούν με τον ΑΒ τρόπο στην πρόκληση. Τι πιστεύετε, το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντέξει 6, 7, 8, 9 μήνες πολιτικού ανταγωνισμού και οικονομικών ταραχών. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σας. Και Διαβάζοντας τους Financial Times φαίνεται ότι το σκάνδαλο Danske είναι και ε, σκάνδαλο της Deutsche Bank. Τι στράβωσε στις υποθέσεις αυτές, Danske και πιθανόν και Deutsche Bank, και τι πρέπει να γίνει τώρα. Τώρα, για τον Ιταλικό τραπεζικό τομέα φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ευαισθησία στις αγορές σχετικά με τους δημοσιονομικούς στόχους των Ιταλών. Υπήρξαν αντιδράσεις που αύξησαν την απόδοση των Ιταλικών ομολόγων και επίσης ε, ε, πλήγησαν και τα κεφάλαια των τραπεζών μέχρι τώρα. Δεν έχει περάσει το πρόβλημα και σε άλλες δικαιοδοσίες, ούτε έφτασε σε ένα επίπεδο όπου αποτελεί σοβαρό πρόβλημα ανησυχίας και για τις τράπεζες. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα φέρει το μέλλον. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσουν οι συζητήσεις και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Προσωπικά νομίζω ότι οι Ιταλικές τράπεζες έκαναν πολλές προσπάθειες για να νοικοκυρέψουν τους, ε, ισολογισμούς, τους να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και θα ήταν πολύ λυπηρό αν πληγούν από τις συνέπειες της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτά τα πράγματα βέβαια συμβαίνουν. Και τα προβλήματα των ελληνικών τραπεζών έτσι άρχισαν από πολιτικές αντιπαραθέσεις. Οπότε ε, ε, ευχόμεθα το καλύτερο. Τι άλλο να πω. Να ελπίζουμε ότι οι Ιταλικές τράπεζες ε, θα βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους, τη φερενκιότητά τους. Γιατί το προσπάθησαν πολύ αυτό και έχουν πετύχει αρκετά. Είχαν καλά αποτελέσματα ε, στο στρες τεστ της τραπεζικής αρχής. Αυτό έχω να πω. Τώρα, ο Όμιλος Ντάνσκε, σχεδόν κάθε μέρα όταν διαβάζουμε τις εφημερίδες, ανακαλύπτουμε καινούριε εξελίξεις. Η Εποπτική Αρχή της Δανίας που είναι η υπεύθυνη και για το ξέπλυμα χρήματος για την καλοσύνη να έρθει στη ποπτικό Συμβούλιο τώρα ήρθε στο, ε, στην Κεντρική Τράπεζα και διαβεβαίωσε και όντως καταβάλει προσπάθειες για να λύσει το πρόβλημα. Ε, υποθέτω ότι τις ίδιες εφημερίδες διαβάζουμε χθες και σήμερα. Δεν θέλω να βλέπω τι τράπεζες του εποπτικού μηχανισμού να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, αλλά συμβαίνει αυτό και είναι και γεγονός είναι ότι δεν ήταν πολλές οι τράπεζες που παρήχαν τέτοιες τραπεζικές υπηρεσίες με ανταποκριτή θα λέγαμε, ανταποκρίτρια τράπεζα στις βαλτικές χώρες. Είναι δύσκολο να παίζει κανείς το ρόλο αυτό της ανταποκρίτριας τράπεζας. Είναι δύσκολο όταν δεν γνωρίζεις τα δεδομένα της χώρας. Ελπίζω να περιοριστεί όσο γίνεται περισσότερο το πρόβλημα. Ε, ας είμαστε αισιόδοξοι, ας ευχηθούμε για το καλύτερο. φαίνεται ότι πολλά ε, κακά ακολουθούν την μη ανεύθυνη τραπεζική πολιτική. Ο Κώστας Μαυρίδης. Thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Νουή, νομίζω ότι θα χρειαστείτε τα ακουστικά σας. Εκτός αν έχετε μάθει ελληνικά. Όχι, οι Γάλλοι δεν είναι καλοί στο να μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Ωραία. Όλα θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω πραγματικά για το έργο που επιτελείτε και σας εύχομαι καλή συνέχεια για ό,τι θα κάνετε. Επειδή είναι και η τελευταία σας παρουσία, ε, δεν θα επικεντρωθώ στα θέματα του ΙΤΙΣ, γιατί αισθάνομαι ότι έχω καλυφθεί. Προσωπικά συμμερίζομαι την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσουμε και με risk neutralization. Τούτου λεχθέντος θα επικεντρωθώ στα NPLs. Αλλά συγκεκριμένα, Μανταμνουή, θα επικεντρωθώ στην περίπτωση της Κύπρου. Από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, μέχρι σήμερα, το δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρου έκλεισε. Αυτό δεν ήταν στις ειδήσει αυτή τη φορά. Αναφέρομαι στο, στο συνεργατικό τραπεζικό ίδρυμα, ξέρετε για ποιο αναφέρομαι, και έκλεισε γιατί μεταξύ άλλων υπήρχαν συσσωρευμένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχω δύο-τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Είχατε ενημερώσει τον Υπουργό Οικονομικών για τα προβλήματα που υπήρχαν σε αυτό το τραπεζικό ίδρυμα. Τον πιέσατε. Είχατε επίγνωση της ανεπάρκειας της διοίκησης που ανέλαβε αυτό το ίδρυμα και διορίστηκαν όλοι πολιτικά. Για να καταλάβετε την ανεπάρκεια τους θα σας πω το εξής. Μέχρι πρόσφατα, μέχρι να καταρρεύσει το Ίδρυμα, θεωρούσαν τους στόκους πάνω στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως κέρδος για το Τραπεζικό Ίδρυμα. Και κρίνοντα εκ του αποτελέσματο, για να κλείσω με αυτό το θέμα, με το συνεργατικό, με το συνεργατικό τραπεζικό ίδρυμα, ε, να σας πω ότι ανέθεσαν τη διαχείριση των FPLs σε μία μόνο εταιρεία, χωρίς διαφανείς διεργασίες αναφέρομαι στην μοίρα. και κρίνοντας εκ του αποτελέσματος έχουμε και εδώ μια τεράστια αποτυχία. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κάπως άσχετο με το θέμα μας. Μαντάμ Νουή, όσοι πιστεύουμε στον ευρωπαϊκό θεσμό, αναμένουμε από τους επόπτες μας να είναι πιεστικοί. Στο, στην Κύπρο γίνονται συστηματικά καταχρήσεις από τις τράπεζες ενάντια στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και αναμένουμε από εσάς, σε αυτό τον τομέα, να συνεχίζετε να παίζετε ένα σημαντικό ρόλο. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, Μία τράπεζα έκλεισε, συγχωνεύτηκε με μια άλλη τράπεζα στη Κύπρο. Δεν μπορώ να σχολιάσω πολλά σχετικά με μεμονωμένες τράπεζες. Μπορώ να σας πω κάποια πράγματα όμως. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για μια τράπεζα που είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν ε, δυσκολίες. Τότε είχε 60% ε, μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μόνο πρόσφατα υποβλήθηκε σε έλεγχο από την ε, Εθνική Τράπεζα της ε, Κύπρου και ζητήθηκε από τον SSM να ε, καλύψει το ρίσκο της εποπτείας. Εξαιτίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων η τράπεζα χρειαζόταν κεφάλαια ε, για την ενίσχυση των αποθεματικών, αλλά και ε, χρειαζόταν και τεχνογνωσία. Ήταν ένας ε, σύνθετο, ήταν ένα σύνθετο ίδρυμα με πολύπλοκες συναλλαγές, ένα δύσκολο περιβάλλον Πράγματι, ε, συζητήσαμε με τις Κυπριακές Αρχές και την Κεντρική Τράπεζα φυσικά, αλλά ε, συζητήσαμε και με τον Υπουργό Οικονομικών. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας με όλους τους Κυπριακούς φορείς, τις Κυπριακές Αρχές. Κατάλαβαν αυτά που ε, λέγαμε ότι όχι μόνο η τράπεζα χρειαζόταν ε, κεφάλαια, αλλά και τραπεζική τεχνογνωσία προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ε, είχε. Και σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης το Σεπτέμβριο του 2017 με στόχο να αποκομίσει και κεφάλαια και τεχνογνωσία. Η ρευστότητα της τράπεζας στο τέλος του 2017 αυξήθηκε ε, ε, ε, αρκετά, ε, εμφανίστηκαν πολλά προβλήματα, ε, έγιναν πολλές δημοσιεύσεις στις κυπριακές εφημερίδες. Αναφέρθηκε τότε και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κύπρου. Όλα αυτά τα θέματα συζητήθηκαν πάρα πολύ. Η διδικασία ιδιωτικοποίησης ε, οδήγησε σε, σε μία πρόταση, ουσιαστικά μία πρόταση, η Hellenic Bank ε, ε, υπέβαλε την καλύτερη πρόταση. νομίζω ότι έχω κρυώσει λόγω της αλλαγή του καιρού. Σας έλεγα λοιπόν ότι η Hellenic Bank έκανε μια καλή πρόταση, έχει καλές δυνατότητες εκτέλεσης. Τώρα έχουμε μία ε, συγχώνευση την Συνεργατική Τράπεζα ε, ε, διαδέχτηκε μια ε, άλλη τράπεζα που υπάγεται στον έλεγχο της Κεντρικής Κυπριακής Τράπεζας. Πιστεύω ότι ότι έχουμε μια ικανοποιητική ε, κατάσταση γιατί ε, δεν είχαμε μια έξοδο από την αγορά χωρίς ε, δεν είχαμε μια έξοδο από την αγορά με σημαντικές επιπτώσεις Τώρα τα NPLs δεν υπάρχουν στο πεζικό ε, εθνικό σύστημα, αλλά τα διαχειρίζεται αυτή η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών ε, στοιχείων και νομίζω ότι ε, το μέλλον διαγράφεται θετικό. Επίσης θετικό είναι ότι η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή με όλους τους φορείς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού παρακολουθούσε ε, το θέμα. Ε, συνεργαστήκαμε και με το Υπουργείο Οικονομικών και με όλες τις Κυπριακές Αρχές. Το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης παρέμενε ενημερωμένο καθ' όλη τη διαδικασία. Δεν έγινε κάποια δήλωση failing or likely to, to fail. Είχατε 9 λεπτά στη διάθεσή σας. Ρώτησα την κυρία Νουή να σχολιάσει και την ε, τις καταχρήσεις των τραπεζών στην Κύπρο. Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας. Αν είχαμε εντοπίσει κάτι θα είχαμε ενημερώσει τις αρχές. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ ε, κυρία Νουή και εγώ σας θαυμάζω για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα και, και όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε μετά τη ε, κρίση. Εγώ δεν θα σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τα δεδομένα, μιας και είναι η τελευταία σας παρουσία εδώ. Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω τη γνώμη σας για κάτι πολύ σημαντικό. Δεν το αναφέραμε μέχρι τώρα και αφορά τον έλεγχο των εποπτικών αρχών. Πριν από κάποιες εβδομάδες αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Επικεφαλών των Εποπτικών Αρχών σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό ε, επίπεδο ε, έκαναν μια, δημοσίευσαν μια ανακοίνωση με Προειδοποίηση σε ό,τι αφορά το, ένα, το λεγόμενο χάσμα ε, εποπτείας. Πράγματι, πολλές αρμοδιότητες πέρασαν στο SSM. Ταυτόχρονα όμως, το ελεγκτικό συμβούλιο ε, έχει ακόμα κάποιες ε, αρμοδιότητες ό,τι αφορά την εποπτεία των ε, τραπεζών. Η κατάσταση είναι αρκετά σύνθετη. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, από την άποψή σας. Πώς βλέπετε τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτό το χάσμα, το εποπτικό, τι μπορεί να γίνει ε, για να βελτιωθεί η ικανότητα των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Και δεύτερη ερώτηση, ε, εδώ και κάποιο καιρό ελπίζουμε να ξεκινήσει ένας διάλογος με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την ε, ε, τροποποίηση της ε, οδηγίας EMID ε, σε ό,τι αφορά το εξή. Θα υπάρξει μία επιτροπή που θα υποβάλει προτάσεις τροποποίησης αν συμφωνεί και το Εποπτικό Συμβούλιο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εσείς είστε υπέρ αυτής της ε, διαδικασίας. Ξέρετε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα και πώς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ για τις δύο ερωτήσεις. Τώρα, η εντολή του ελεγκτικού συνεδρίου που θα μπορούσε να έχει κενά. Στην ΕΚΤ ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν ε, μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Οι, κρατικοί, οι δημόσιοι ελεγκτές ε, περιορίζονται στο έργο τους από πολλές δικαιοδοσίες. Σε άλλες η εντολή του δημοσίου ελεγκτή περιορίζεται στον έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης των δημοσίων ε, κεφαλαίων που έχουν ληφθεί. Επίσης, η Εθνική Αρμόδια Αρχή ε, φροντίζει για την εφαρμογή της νομοθεσία που προβλέπει δυνατότητα, αλλά όχι υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να ζητήσουν δημοσίευση ε, πληροφοριών και κοινοποίηση στο ελεγκτικό συνέδριο. Ε, η άποψη της τράπεζας, της κεντρικής τράπεζας, είναι ότι αυτό δεν είναι σωστό. Κατά τα άλλα, εμείς παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τις απαραίτητες πληροφορίες για να δουν την ε, λειτουργία της τράπεζας, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό είναι καινούριο για το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά και πάλι εμείς δώσαμε στο ελεγκτικό συνεδρίο όλες τις πληροφορίες. Και δεν νομίζω ότι είναι θεμητό ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να παραπονείται όταν, παίρνει όταν δεν παίρνει πληροφορίες που είναι εκτός ε, πεδίου εντολής. Τώρα για το ΙΜΙΡ 2 είναι σωστό ότι στα πλαίσια του Brexit η έγκαιρη ε, έγκριση του ΙΜΙΡ και η τροπολογία στο άρθρο 22 θα διασφαλίσει ότι οι, ευρωπαϊκές, οι αρχές θα έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσει ε, ενδεχόμενους ε, κινδύνους ε, μετά τον Brexit. Ναι, και η διαδικασία μη ένστασης που είπατε ότι είναι... Α, δεν το ανέφερα αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς λειτουργεί σε άλλα ιδρύματα, σε άλλα θεσμικά όργανα. Θα έλεγα γενικά ναι, αλλά δεν είναι και εγγύηση ότι είναι ε, ο καλύτερος τρόπος αυτός. Θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό με τα λόγου γνώσεως. Υπερβάνς Περέζ. Ναι, τελικά δεν μιλήσαμε και πολύ για το Brexit. Είναι φυσικό γιατί δεν είστε υπεύθυνοι για την ε, εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά, Ωστόσο, ε, μέσα στην προοπτική αυτού του διαζυγίου, εσεί δεν ανησυχείτε μήπω τελικά ε, αυτό που είπατε ότι ο τραπέζικό τομέα θα πάει καλύτερα, είναι πιο ανθεκτικό, αλλά ένα κομμάτι του τραπεζικού τομέα δεν μα απασχόλησε και τόσο. Είναι η σκιώδης τραπεζική και αυτό το σύστημα. Εκεί σε αυτή την αξιολόγηση δεν προέβημεν. Πρόσφατα είπατε ότι είχατε αμφισβητήσεις για το θέμα αυτό, ότι υπήρχε δηλαδή περιθώριο ε, προόδου όσον αφορά την κερδοφορία των τραπεζών. Την τελευταία θητεία είχαμε ασχοληθεί με μια πρώτη, πρόταση που λεγόταν BSR, ε, Πώς λοιπόν θα καλύψουμε το θέμα της τραπεζικής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. Γιατί το βλέπουμε καλά. Αν δούμε ένα μοντέλο τραπεζικό το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε μια χώρα ε, μόνο και έχουμε ε, διαφορετικό στη διπλανή, δεν προχωράει καλά το πράγμα. Τρίτη ερώτηση. Είδαμε στην υπόθεση Banco Popular και ήταν η εντύπωση που είχαμε ότι σε περίπτωση εξυγίανσης ή ε, failing ή likely to fail κατάσταση της το θέμα της διαβίβασης των πληροφοριών ανάμεσα στο δικό σας ε, θεσμό και εκείνον που προεδρεύει ο Ελκ Κένιγκ και εκεί υπάρχει περιθώριο προόδου. Εσείς αυτά όλα πώς τα αναλύετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης τραπεζική, ναι βεβαίως ε, και μας προβληματίζει για το ότι υπάρχουν τραπεζοειδείς δραστηριότητε που δεν είναι υπό απόλυτο έλεγχο και μπορεί να έχει αυτό επιρροή ε, που θα λειτουργήσει αλυσιδωτά. Εμείς έχουμε δει το, έχουμε το, shadow, το shadow banking, τη τραπεζική, αλλά δεν έχει υπάρξει πρόοδος και δυστυχώς αυτό είναι κρίμα βεβαίως. Ε, έγιναν πρόσφατα δηλώσεις από τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ για το γεγονός ότι ανησυχούσε για τα διάφορα ε, ταμεία, την κατάσταση των ταμείων και κάποιων από αυτά. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Ε, εκείνος είναι υπεύθυνο για την δημοσιονομική σταθερότητα, για το κοινό όφελος και την νομισματική πολιτική και το SSM και θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η ΕΚΤ. Τι σημαίνει εκείνο το BSR είναι το Banking Structure Review για το διαχωρισμό, για τη μεταρρύθμιση. Ναι. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην ε, Ευρώπη. Ε, ναι. Χρηματιστήρια, ναι. Γιατί όχι να υπάρχει παραδοσιακή εμπορική τράπεζα από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά οι, οι υπόλοιπε δραστηριότητε των τραπεζών. Αυτό θα ήταν πολύ απλό, αλλά στην Ευρώπη η οικονομία χρηματοδοτείται βασικά από τις τράπεζες 70% και για την χρηματοδότηση των ε, μεγάλων τροπεζών. Εκείνες παίζουν τεράστιο ρόλο στη λειτουργία της αγοράς και είναι εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση, αν όχι αδύνατον το να το καταφέρουμε. Εάν κάνουμε market making με το proprietary trading, έχεις πρόβλημα με την οικονομία. Αν το βάλεις με τις παραδοσιακές εμπορικές τράπεζες, ε, έχεις πολύ λίγα να ξεχωρίσεις και να διαχωρίσεις. Το είδα στη χώρα μου, ξεκινώντας από την βούληση μιας νέας πολιτικής ομάδας να κάνει κάτι πολύ αυστηρό, ε, όσο προχωρούσε η υπόθεση τα αρνητικά στοιχεία ήταν πιο πολλά από τα θετικά. Και η Γερμανία και η Γαλλία προέβησαν σε μεταρρυθμίσεις λογικές όπου πρέπει να φτάσει κανείς σε ένα επίπεδο proprietary trading για να μπορέσει να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό. Και το market making είναι σε ένα τελείως άλλο επίπεδο. Διαφορετικά δεν είμαι βεβαία πώς μπορεί αυτό να γίνει στην πράξη. Επιπλέον, ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι τράπεζες για περίπλοκες συναλλαγές για ίδιους λογαριασμούς είναι ε, ε, πολύ μικρότερος, πολύ χαμηλότερος, έχει μειωθεί. Θα επανέλθει το θέμα σίγουρα, ε, ειδικά όταν η κερδοφορία είναι χαμηλή, θα επανέλθει. Για την ώρα όμως δεν μας απασχολεί το θέμα. Η συνεργασία με την με την SIB Είμαστε μέλη, είμαστε παρατηρητές, πάντως είμαστε μέσα στο, στο Συμβούλιο του SRB, ενώ η Κένιγκ δεν έχει ε, θέση στο Εποπτικό Συμβούλιο. Δώστε της μια θέση. Κάτι όμως που μπορεί το SRB να ρωτήσει κάποιες φορές που δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν είναι δική μας υπόθεση, γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε, ε, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ε, θα δούμε όταν θα αρχίσουν να χάνουν τη δύναμή τους οι τράπεζες. Ε, τότε θα δούμε τον κίνδυνο. Θα ήταν πιο άνετο βέβαια να τα έχουμε κάνει όλα εκ των προτέρων, ίσως. αλλά δεν το κάνουμε γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και βλαβερό. Μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν κάποιες αδυναμίες σε κάποια σημεία να, να φτιάχνουμε αποφάσεις ε, ε likely to fail. Όταν είμαστε σε μια κατάσταση ανάλογη μπορεί να ξεκινήσουμε και να σκεφτόμαστε πως ίσως το χρειαζόμαστε. Εν γέννη ε, συζητούμε με την Έλκη Κένιγκ πριν να το συζητήσουμε με το ε, στους ανθρώπους του Συμβουλίου ε, ακριβώς για να μην είναι πολλοί ε, που γνωρίζουν το, το πρόβλημα. Πάντως ε, μοιραζόμαστε πολλά, έχουμε συνεργασία, έχουμε την αναθεώρηση του Μνημονίου Συνεννόησης και να προσθέσω ότι όταν έχουμε ε, ε, στάσεις κρίσης όλοι συνεργάζονται πάρα πολύ καλά και πάντα διότι γνωρίζουμε πως είναι κάτι σοβαρό, ότι, ότι δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος. Ότι η διαδικασία πρέπει να είναι αλάνθαστη και όλοι πρέπει να έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσουμε να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Πέρα από το να δοθεί θέση στην ΕΛΚΕ στο SSM, πράγμα το οποίο υποστηρίζω στεναρά, δεν βλέπω κάτι άλλο, κάποια, άλλη δυνατότητα. Ευχαριστώ. Η Ντανούτα Χούμπνερ. Κυρία Νοή, ίσως θα θυμάστε ότι στη διάρκεια της θητείας σας μέγα θέμα ήταν οι εθνικές επιλογές και η ε, διακριτική ευχέρεια και συχνά αναφερθήκατε σε αυτή την πρόκληση για τη δικιά σας εργασία. Επίσης βλέπουμε πως υπάρχει απόκληση ανάμεσα στα κράτη-μέλη στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τους κανονισμούς, στον τρόπο με τον οποίο μεταγράφουν τις οδηγίες στην εθνικό τους δίκαιο στους διάφορους τομείς. Επίσης διαπιστώνουμε πως οι εθνικοί επόπτες συχνά εξετάζουν το ίδιο θέμα αλλά αντιδρούν διαφορετικά. Υπάρχει και αυτού του είδους η απόκληση και η ποικιλομορφία που προκύπτει από τις εθνικές εποπτικές αρχές και τη διακριτική ευχαίρεια που έχουν αυτές. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι είδους συστάσεις θα κάνατε στον διάδοχό σας Τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε αυτού του είδους τις αποκλήσεις που προέρχονται από διάφορους τομείς. Προηγουμένως μιλήσατε για τον κατακαιρματισμό εν γέννη που εξακολουθεί να ισχύει στην Ευρώπη και νομίζω πως αυτού του είδους οι αποκλήσεις συμβάλλουν σε αυτό. Τι είδους προσπάθειες λοιπόν μπορούν να γίνουν στην Ευρώπη για να περιοριστεί αυτό το πρόβλημα. Εθνικές επιλογές. δεν μπορούν να εξαφανιστούν τελείως οι εθνικές διαφορές. Αναρμονίζουμε την εφαρμογή στον ενιαίο μηχανισμό ε, εποπτείας. Αυτό είναι ήδη σημαντικό, να έχουμε δηλαδή ισότιμο πεδίο για όλους μέσα στο συγκεκριμένο πεδίο ε, του κανονισμού. Ε, Έχουμε εναρμονίσει τα πάντα εκτός από το συμβιβαστική της Δανίας για την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εταιριών. Δυστυχώς, για άλλα πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί αυτά εξαρτώνται από τους εθνικούς νομοθέτες. Η συμβουλή μου, αν τη δεχτείτε, θα ήταν να τους δώσετε στις εθνικές αρμόδιες αρχές αντί για τους νομοθέτες, δηλαδή τις εθνικές εποπτικές αρχές, δηλαδή το SSM για τις χώρες γιατί έτσι θα είχαμε έναν μόνο τρόπο να ασκούμε τις εθνικές επιλογές μέσα στο πλαίσιο του ενιαίου μηχανισμού ε, και θα είχαμε όπως είπα ισότιμο πεδίο. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα ήταν αυτός ο τρόπος. Ελπίζω εγώ σε υπόπτυση ότι θα ήταν ο πιο αυστηρός τρόπος εφαρμογής αλλά εν πάση περιπτώσει θα δεχτώ ότι αποφασίσουν τα μέλη του ε, Συμβουλίου. Ήδη τον έχουν οι εθνικές εποπτικές αρχές ε, την αρμοδιότητα για την εφαρμογή αυτών των μέτρων θα ήταν πολύ σημαντικό αντί να την έχουν την ευθύνη οι εθνικοί νομοθέτες. Ήδη για τις εξαιρέσεις ε, τα waivers έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε ε, την άδεια για ρευστότητα μέσα σε μια ομάδα ανάμεσα στις κρυμμένες τράπεζες. Αλλά είναι σχεδόν άχρηστο γιατί είναι σταγόνα στον ωκεανό στην ουσία λόγω του μεγάλου ορίου έκθεσης η άδεια για μεγάλη δυνατότητα έκθεσης είναι στα χέρια του εθνικού νομοθέτη. Οπότε προφανώς αν μια ομάδα είναι έτοιμη να δώσει στήριξη ρευστότητας ενδο, μέσα σε ομάδες εντός του ε, SSM, ε, τότε σημαίνει ότι η ρευστότητα δεν βοηθάει και πολύ. Διασυνοριακή αφεργιότητα δεν υπάρχει, ετέθη επιτάπητος, αλλά δεν ε, έγινε δεκτό. Ήδη η μεγάλη, ε, τα μεγάλα ανοίγματα ε, τελειώνουν αν η ρευστότητα υπάρχει ε, και όπως σας είπα αυτό είναι που χρειάζεται. Κάτι άλλο ξέχασα? Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ευκαιρία. Να έσω μία ερώτηση. Γιατί βλέπω τον ε, πιθανό σας διάδοχο εδώ ήδη. Εσείς ήδη αναφέρατε πολύ καλές ε, πιθανότητες, μάλλον θέματα ως ε, επιπλέον ατζέντα ή επιπλέον συστάσεις που θα δώσετε στο διάδοχό σας για τη διαχείριση αυτού του πολύπλοκου μηχανισμού που είναι το OSSM. Επίσης, η Κάνατε ένα σχόλιο με το οποίο είμαι απόλυτα σύμφωνος και όσον αφορά την κατάσταση των spread ε, και των ομολόγων στην Ιταλία, αυτό μας κάνει όλους να ανησυχούμε. Και βεβαίως μια μακρά περίοδος υψηλών spread δεν είναι βιώσιμη. Όλοι λοιπόν ευχόμαστε το καλύτερο Ευχαριστήσω λοιπόν για την καλή σας εργασία και για το input στο SSM όσον αφορά τους κινδύνους και την, την ε, κεφαλαϊκές απαιτήσει. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο διάδοχος ε, πρέπει να εφαρμόσει τις καλύτερες εποπτικές πρακτικές και στην Ευρώπη και αλλού για το ε, Συμβούλιο Εξυγίανσης συνεργασία με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ε, η Κομισιόν, ο SRB, εμείς είμαστε αδελφά όργανα ε, με δέσμευση υπέρ των ιδεοδών της Ένωσης και έχω, έχω ε, σίγουρα στη βαρότητα, στην προσέγγιση των τραπεζών. Πολλές φορές ε, είναι ε, αναγκαίο να είμαστε αρκετά ισχυροί για να περάσουμε τις απόψεις μας και σίγουρα επιμονή γιατί η δουλειά είναι πολύ Αλλά ξέρω ότι ο Ανδρέα είναι, εργάζεται σκληρά για τις Ιταλικές τράπεζες. Είμαι ευτυχής διότι ε, συνέβαλαν σε μια βελτίωση της κατάστασης. Δεν έχουμε δει αρνητικές επιπτώσεις ούτε ε, έμεσες ε, επιπτώσεις σε άλλες χώρες. Ελπίζω να μείνουμε εκεί γιατί θα ήταν πολύ κακό να ανατρέπονται οι προσπάθειες που έγιναν και τα καλά αποτελέσματα να αναστρέφονται. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Το εύχομαι πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ όλες οι ομάδες και όλοι οι ομιλητές Ντανιέλ σε συνεχάρισαν όπως είδε και σε συνεχάρισαν για την δουλειά σου, σε ευχαρίστησαν. Ε, ε αξίζεις το χειροκρότημα, το είπα και στην αρχή και ήθελα να το επαναλάβω με θέρμη και στο τέλος. Εκτιμούμε πάρα πολύ όσα έκανες. Έγραψες ιστορία στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση γιατί η δημιουργία του SSM ήταν καταπληκτικό έργο και η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που θα γράφει στα βιβλία της ιστορίας. Θα κριθούμε στο μέλλον με βάση αυτά που κάναμε και νομίζω ότι όλη η ομάδα ήταν εξαιρετική. Ευχαριστούμε γι' αυτό και ευχαριστούμε και για την άρεστη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πάντα ήταν θετικότατη, αποτελεσματική και όταν είχαμε διαφωνίες πάντα η συζήτηση ήταν επικοδομητική γιατί αυτός είναι καλός τρόπος ε, να ε, ενημερώνεται και το κοινοβούλιο ε, που πρέπει να παρακολουθεί τα θέματα λογοδοσίας. Ελπίζω και στο μέλλον υπάρχει η διαφοσίωση και σεβασμός προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μεταβιβάσω τα καλά σας λόγια ε, στο προσωπικό, στην Φραγκφούρτη και στις εθνικές αρμόδιες αρχές. Δύο λεπτά διακοπή και συνεχίζουμε με την ακρόαση. let's start this new point in Επόμενο θέμα. Δημόσια κρόαση με τον προτινόμενο υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Υποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Έχουμε μια συνέχεια στη μερίσια διάταξη. Ε, είχαμε την κυρία Νουή, τον κύριο Ανρία τώρα, τον Ενρία, τον καλωσορίζω. Στις 7 Νοεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, έχοντας λάβει τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου, πρότεινε τον κύριο Ανδρέα Ενρία ως διάδοχο της κυρίας Νουή ως πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ από την 1η Ιανουαρίου του 2019 για διάρκεια θητείας πενταετή. Ε, να καλωσορίσω τον κύριο Ενρία, ο οποίος ε, ε, τώρα είναι, όπως γνωρίζομαι, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τον κανονισμό SSM, το Συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του ΙΣΕΚΤ μεταξύ προσωπικότητων εγνωσμένου κύρους και πείρα σε χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα με βάση διαδικασία ανοιχτής επιλογής μετά από πρόταση της ΕΚΤ και μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. η επίσημη αυτή ακρόαση δημοσία είναι πολύ σημαντική για την λογοδοσία του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου υπογραμμίζει την ε, λογοδοσία του Προέδρου. Το Κοινοβούλιο συμμετείχε άτυπα και στις προηγούμενες ε, διαδικασίες. Ευχαριστώ τον κύριο Ενρία και όλους τους υποψήφιους, τους υπολείπους που όλοι ήταν ε, υψηλής ε, περιοπής. Και τώρα θα ακούσω με τον κύριο Ενρία. Σας δίνω το λόγο για την, ε, τις αγωγικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζω ευχαριστώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και τους συντονιστές της ΕΚΟΝ που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής ε, με πρότειναν. Ήταν μεγάλη μου τιμή να δω, να, προτι... Ε, να προτείνομαι ανάμεσα σε πολλούς άλλους άξιους υποψηφίους. Ποια είναι οι βασικές προτεραιότητες στα επόμενα πέντε χρόνια. Πρώτον, ολοκλήρωση του ξεκαθαρίσματο ε, ξεκαθαρίσματος των ισολογισμών των τραπεζών. Οι εποπτικές πολιτικές θα πρέπει να ασκήσουν πιέσει σε κάθε τράπεζα χωριστά για να ε, προσαρμοστούν γρήγορα. Όσο γρήγορα τελειώσουν οι τράπεζες με τους παλιούς κινδύνους, τόσο καλύτερα για την πραγματική οικονομία ολοκλήρωση και επιμερισμός κινδύνου. Μετά την αρχή της κρίσης, ο τραπεζικός τομέας ε, έδρασε ως επιταχυντής της ε, ε, κρίσης. Ο ιδιωτικός επιμερισμός κινδύνου δεν ήταν αρκετός. Θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία παντού στα κράτη-μέλη σε όλες τις τράπεζες σύμφωνα με τον κανονισμό SSM. Συνολική δράση χρειάζεται από όλους τους πολιτικούς ώστε η Τραπεζική, σύστημη, η Τραπεζική Ένωση να γίνει πραγματικότητα. Η πρόθεση της ολοκλήρωσης και το ξεκαθάρισμα των ισολογισμών ε, είναι απαραίτητες αλλά και υπαρξιακές προκλήσεις. Η Τραπεζική Ένωση δεν θα επιβιώσει αν μας πιάσει η επόμενη κρίση να ασχολούμεθα με την κακιά κληρονομιά της παλιάς κρίσης ή με κατακαιρματισμένες εθνικές πολιτικές. Ε, θα πρέπει να δούμε τη χρηματοδότηση και το ε, κίνδυνο. Ε, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ και πρέπει να δούμε και τις πρακτικές αξιολόγησεις οι τράπεζες ε, του, της ε, ε, Ένωσης πολλές φορές δεν ε, αντιμετωπίζονται με θετικό τρόπο, δηλαδή δεν θεωρούνται όλες ελκυστικές. Τέλος, το θέμα της διακυβέρνησης και της κουλτούρας θα του κινδύνου θα πρέπει να συνεχιστούν. Θα πρέπει να έχουμε δια... διασφαλίσεις τέτοιες που να ε... ισχύουν για όλο τον τραπεζικό χώρο. Οι επόπτες ε, συμβάλλουν επίσης στην μείωση των ε, σκανδάλων λόγω ξεπλήματος. Ε, ο επόπτης παρουσιάζεται ως αυστηρός. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των εποπτικών δράσεων από την πείρα μου στην ε, τραπεζική αρχή πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί ισορροπία μεταξύ ανάγκης για εμπιστευτικότητα αλλά και από την άλλη ανάγκη για δημοκρατική λογοδοσία που επιτρέπει επαρκή έλεγχο. Ε, προς τη βιομηχανία καλή ισορροπία μπορεί να βρεθεί μεταξύ του θεμητού εποπτικού στόχου που όμως ε, θα αποφεύγει μηχανιστικές προσεγγίσεις και την ανάγκη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του επόπτη να γίνει εύληπτο για τις τράπεζες και, ε, για τις επιχειρήσεις, Το βάρος των ζημιών σε περίπτωση κρίσης ε, κυρίως το επομίζονται οι ιδιώτες επενδυτές. Πρέπει γι' αυτό να είναι πιο διαφανές. Ξέρω ότι είναι αντιφατικό αυτό στην εποπτική κοινότητα, αλλά είμαι πεπισμένος ότι τα μαξιλάρια προστασίας είναι χρήσιμα. Επίσης, ε, είναι ε, πολύ σημαντικό και το πρόγραμμα αξιολόγησης της σταθερότητας. Πρέπει να ε, εντοπίσει τον κίνδυνο που δέχονται να αναλάβουν οι τράπεζες. Εμείς λίγο πιο, λίγο πιο αργά για τη διερμηνία. Η, η πτώχευση της τράπεζας δεν είναι αποτυχία του επόπτη ε, κατά ανάγκη. Ε, η δημιουργία της εποπτείας άρχισε στην Ευρώπη ε, πριν από πολλά χρόνια. Εγώ ήμουν και στον τραπεζικό χώρο μέχρι που έφτασα στην τραπεζική αρχή. Είμαι ανεξάρτητος από την βιομηχανία, τις εθνικές αρχές, τους πολιτικούς. Επίσης έχω μια μέθοδο εργασίας που στηρίζεται στην ειλικρίνεια, τη διαφάνεια και στον εκτενή διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους. Έχω καλές εσωτερικές επικοινωνίες με το προσωπικό. Ε, είμαι διατεθειμένος να αναλάβω ευθύνες κάτω από δύσκολες συνθήκες και όταν ο οργανισμός δεν είναι σαφώς υποχρεωμένος να δράσει. Ε, βλέπω τον εαυτό μου και ελπίζω έτσι να με βλέπετε ως έναν δημόσιο λειτουργό σε ενωσιακό επίπεδο. Αν ε, με διορίσετε, οι αξίες αυτές θα διέπουν την δράση μου. Ε, θα ε, έχω την τύχη να συνεχίσω τα καλά αποτελέσματα της προκατόχου μου, της κυρίας Νουή, με την οποία συνεργάστηκα πολλές φορές στη σταδιοδρομία μου. Η ποιότητα των θεσμών εξαρτάται από το, τους ανθρώπους που τις τελεχώνουν. Ε, είχα τη δυνατότητα από πρώτο χέρι να δω το εποπτικό προσωπικό και την υψηλή ποιότητα της δουλειάς τους ο SSM δεν θα μπορούσε να ε, λειτουργήσει χωρίς την αφοσίωση και το προσωπικό από τις εθνικές αρχές και τις εποπτικές ομάδες και την, ε, εποπτική, την εποπτεία ε, όλων των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, προβλέψαμε μόνο πέντε λεπτά για τη δική σας ομιλία. Θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι από ε, την Τανιάλα Χούμπνερ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για το κρατικό χρέος. Θα ήθελα να σα ρωτήσω για την άποψή σας σχετικά με τις ε, αλλαγές ρυθμίσει, στις ε, ρυθμίσεις για τη διαχείριση του κρατικού ε, χρέους. Κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνουν κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο του SRB και συζητείται η δημιουργία ενός οργανισμού διαχείρισης των περιουσιακών ε, στοιχείων. Εσείς τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Ποια μπορεί να είναι η συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Αρχών για τη ε, διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Τι μπορεί να γίνει ε, σε αυτά τα πλαίσια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ε, πρόσφατα ε, ή μάλλον πριν από κάποια χρόνια δημοσίευσα τη γνώμη μου σχετικά με αυτά τα θέματα. Εμένα η, εμπειρία μου μου έχει διδάξει κάποια πράγματα σχετικά με ε, ε, τα κρατικά ομόλογα. Πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητη η διαφάνεια. Στην αρχή ε, δεν ήταν καταπνοητό το ε, ποια κρατικά ομόλογα διέθεταν οι τράπεζες και ποια ήταν η έκθεσή τους στο, στο κρατικό χρέος. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Ζητήσαμε από τις τράπεζες ε, να ε, ε, έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο κεφαλαίων, αποθεμάτων. Πιστεύω πως για να λειτουργήσουν αυτά τα αποθέματα προστατευτικά σε περίπτωση κρίσης πρέπει να ε, μπορούν οι τράπεζες να τα ρευστοποιήσουν ε, εύκολα άμα το χρειαστούν. Και κατά τη γνώμη μου είναι και αυτό πολύ σημαντικό για τη θέσπιση της ε, απαραίτητης πειθαρχίας, κάτι που δεν έγινε με την κρίση στο παρελθόν. Το επίπεδο συγκέντρωσης είναι ένα επίσης σημαντικό θέμα. Είδαμε ένα σημαντικό επίπεδο συγκέντρωσης των κρατικών ομολόγων. Σε λίγες μέρες κάποιες ε, τράπεζες ε, είχαν 8 ε, με 9 φορές το Tier 1 κεφάλαιο υπομορφή κρατικών ομολόγων. Η πρότασή μας ήταν να υπάρχει μια μικρή επιβάρυνση στο κεφάλαιο που να ξεκινάει από η οποία θα ε, αυξάνεται σταδιακά ανάλογα με τη συγκέντρωση των κρατικών ομολόγων. Αυτή ήταν η άποψή μου, αλλά αυτό αφορά ε, τη ρύθμιση και όχι την εποπτεία. Πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση φυσικά και είναι ε, σημαντικό που δεξιάγεται αυτή η συζήτηση. Ε, χρειάζονται ίσοι όροι ε, ανταγωνισμού και επιτελείται πολύ σημαντικό έργο εδώ. Πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη και την ευρωπαϊκή οπτική γωνία. Εγώ είμαι υπέρ ε, της πρότασης που δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την οποία πρέπει να υπάρχουν ε, ασφαλή περιουσιακά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αντιδράσεις όμως σε αυτή την πρόταση ήταν αρκετά αρνητικές μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Περές, ε, καλησπέρα σας. Πριν από λίγες μέρες μιλήσατε για το συντονισμό των τεστ αντοχής και των εποπτικών δράσεων. Ε, έχετε εμπειρία σε αυτό το τομέα και θα συνεχίζετε να έχετε στα πλαίσια των μελλοντικών καθηκόντων σας ως ε, Συν εισηγητής, ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα υποστηρίξετε την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ποια είναι η γνώμη σας για το συντονισμό των αρμοδιοτήτων του ε, ε, SSM και των άλλων αρχών προκειμένου να είναι επιτυχή τα τεστ αντοχής. Η προκάτοχό σας ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσεχώς θα δημοσίευε την άποψή σας σχετικά με τη νέα πρόταση της Κομισιόν για την, το ξέπλυμα χρήματος ε, η γνώμη σα, ποια θα ήταν σχετικά με αυτό το θέμα και ε, κατά τη γνώμη σα, ποιο θα έπρεπε να είναι το χρονοδιάγραμμα προκειμένου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να υποβάλει την ε, άποψή σα. Φυσικά ξέρω ότι, δεν, ε, ότι είστε του SSM, πρέπει όμως να προχωρήσουμε γρήγορα και άμα καθυστερήσει η άποψη τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, θα είναι πια πολύ αργά. Ευχαριστώ πολύ για το stress test και τις εποπτικές δράσεις. Πρέπει να πω πρώτα απ' όλα ότι υπήρξε κάποια δυσκολία στην αρχή στη σχέση μεταξύ τραπεζικής αρχής και ΕΚΤΕ. Εμείς ε, είχαμε το εποπτική, εποπτικά καθήκοντα και η ΕΚΤΕ επίσης, οπότε ήταν δύσκολο να ε, βρούμε ε, μια λύση. Αλλά στους δύο ε, επόμενους γύρους αυτού του εγχειρήματο προχωρήσαμε καλά και όλο και βελτιωνόταν η συνεργασία μας σε επίπεδο προσωπικού. Επιτελικό. Τώρα, στην περίπτωση που αναφέρατε, νομίζω ότι Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα σύστημα λειτουργικό που δίνει αποτελέσματα, αλλά είναι λίγο ε, βαρύ, επαχθές, ε, δεν ικανοποιεί όλους. Και η Ντανιέλ Νουίγη είπε χθε σε μια διάσκεψη ότι το εγχείρημα είναι πολύ βαρύ για την ε, ΕΚΤ ως εποπτικό μηχανισμό. Τώρα Έχουμε ένα εγχείρημα το οποίο γίνεται σε δύο δόσεις αν θέλετε. Το πρώτο είναι η πλευρά της τραπεζικής αρχής που επικεντρώνει την συγκρισιμότητα και δημοσιεύει τα αποτελέσματα και μετά έχουμε την εποπτική αξιολόγηση που γίνεται μετά και που σε κάποιες χώρες δημοσιεύεται, σε άλλες τα αποτελέσματα δεν δημοσιεύονται καν. Οπότε οι προτάσεις αποσκοπούν στο να βελτιωθεί ε, και να εξατομικευθεί η εποπτική εργασία χρήσιμη για τους επόπτες και το κομμάτι της τραπεζικής αρχής πρέπει να γίνει λίγο πιο ε, αποτελεσματικό ε, σε γενικότερο επίπεδο με εργαλεία από πάνω προς τα κάτω. Εγώ θέλω να αρχίσει μια συζήτηση και θα δούμε τι θα πούν και οι συνεργάτες και στην ΕΚΤ και το προσωπικό. Ε, είναι καλό να ε, υπάρχουν ε, καλά ρυθμισμένες σχέσεις μεταξύ των δύο αρχών η τραπεζική αρχή πιο γενικά και η εκτέ εξατομικεύει τα στρες test στις πραγματικότητες της κάθε τράπεζας και προχωρεί σε βάση κατά τράπεζα. Εμείς συμμετείχαμε στην ε, ομάδα προβληματισμού της Κομισιόν και εγώ προσωπικά συμφωνώ πολύ με τα, συμπεράσματα. Μακροπρόθεσμα χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σύστημα για την καταπολέμηση του ξεπλήματος. Μάλλον για κανονισμό πρέπει να πάμε λοιπόν παρά οδηγία άμεσα εφαρμόσιμο κανονισμό με λεπτομερείς κανόνες και την αποκέντρωση των ε, αρμοδιοτήτων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Οπότε οι προσωρινές λύσεις που θα προσπαθήσουμε να ε, ε, κάνουμε είναι επανεξέταση σαφής και αναθεώρηση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα ε, σαφής συνεργασία και συντονισμός μεταξύ όλων των εποπτών και των προληπτών των προληπτικών μηχανισμών και κοινή κατανόηση του πώς θα πρέπει να ενταχθεί η καταπολέμηση του ξεπλήματος στους προληπτικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Ωραία. Ραμόν Τρεμόζα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Ενρία. Ελπίζω να σας ψηφίσει το Κοινοβούλιο και να διοριστείτε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο τα επόμενα χρόνια. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, για τον Banco Ποβουλάρ. πριν από 1,5 χρόνο είχαμε το πρόβλημα. Τι διδάγματα αντλήσαμε όλοι μαζί. Η ΕΚΤ τώρα παίζει το ρόλο του Ευρωπαίου δημοσιονομικού επόπτη. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα. Δεν αναζητώ ευθύνες εδώ, απλώς πολλοί στην Ισπανία ανησυχούν, έγιναν προσφυγές. Τι πιστεύετε ότι ε, φαίνεται από όλη αυτή την ιστορία, πώς θα χειριστούμε άλλες ενδεχομένως. Και δεύτερη ερώτηση για την Ιταλία. Γιατί έχουμε τώρα το θέμα του δημόσιου χρέους, του ελλείμματος, συγγνώμη. Η Ιταλία είναι η μόνη χώρα όμως που τα τελευταία 20 χρόνια είχε δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μεγάλο στα 19 από τα 20 τελευταία χρόνια. Ε, το θέμα είναι το κόστος του δημοσίου ελλείμματος, ε, ε, επιτόκια κλπ. Θα μπορούσε ο ESM να βοηθήσει την Ιταλία να επαναχρηματοδοτήσει το Ιταλικό δημόσιο χρέος και να μειώσει το ποσό δηλαδή τα Ιταλικά χρήματα των φορολογουμένων, τα χρήματα των Ιταλών φορολογουμένων θα μπορέσουν έτσι να χρησιμοποιηθούν για μεταρρυθμίσεις ε, και άλλα χρήσιμα μέτρα. Ε, μα δεν θα τον βάλουμε επικεφαλής του ESM τον κύριο Ενρία. Αλλά βέβαια δεν πειράζει, δεν θα τον εμποδίσω να απαντήσει. Για τα διδάγματα από την Banco Popular, πολλά διδάγματα υπάρχουν βέβαια. Είχαμε την τύχη στις πρώτες περιπτώσεις να χρησιμοποιήσουμε τα καινούργια εργαλεία ε, από την σχετική οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών και την ανάκαμψη γιατί θυμάμαι ότι υπήρχαν πολλές ανησυχίες που είχαν εκφραστεί στο παρελθόν σχετικά με την ικανότητά μας να διαχειριστούμε ένα τέτοιο σύνθετο σύστημα με λήψη αποφάσεων σε πολλές αρχές, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ως ένα βαθμό πρέπει να ε, τον SSM που μίλησε για ε, αποφάσεις σχετικά με τους, τα ιδρύματα που μπορεί να πτωχεύσουν ή διατρέχουν, πτωχεύουν ή διατρέχουν τον κίνδυνο να πτωχεύσουν. Η, συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα και με την Κομισιόν λειτουργήσε πολύ καλά προκειμένου. Όλοι είπαν ότι ένα από τα βασικά σημεία που ανέδειξε η υπόθεση Banco Popular είναι η σημασία της ρευστότητα και της εξυγίανσης. Αν εξυγιάνεται την τράπεζα πρέπει να παρέχεται ρευστότητα από την πρώτη μέρα μόλις ξαναγυρίσει στην αγορά η τράπεζα. Και δυστυχώς, και αν θυμάμαι καλά, η Banco Popular είχε 17 δις ανάγκες ρευστότητα στις πρώτες μέρες μετά την εξυγίανση Υπήρχε λοιπόν ένας ισχυρός αγοραστής και μόνο αυτό ε, αντιμετώπιζε το, το θέμα της ρευστότητας. Ε, και στη ΣΥΠΑ υπάρχει παρόμοιος μηχανισμός και στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέχονται, ε, παρέχεται ρευστότητα. Ε, αυτό δεν το έχουμε όμως ε, λύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το λύσουμε. Επίσης, το γεγον... έχουμε πολλές τράπεζες που ε, στηρίζονται στο bail-in. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνουμε bail-in και μετά τη Δευτέρα μπορεί να ξαναλειτουργήσει η τράπεζα. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο ε, είναι ε, το πρόβλημα. Και αυτό που είπατε, ότι έχουν γίνει πολλές προσφυγές σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι το θέμα το, της αποτίμησης πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Καμιά φορά οι τράπεζες δεν έχουν αρκετά ε, υψηλής ποιότητας δεδομένα, ούτως ώστε οι αρχές εξυγίανση να κάνουν καλή αποτίμηση σε συμπιεσμένο χρονικό διάστημα. Η σωστή πληροφόρηση πρέπει να υπάρχει και θα πρέπει ο μηχανισμός της αποτίμησης ε, να λειτουργεί καλά. Για την Ιταλία δεν μπορώ να πω για τα δημοσιονομικά, σίγουρα δεν, είναι, δεν συμφωνώ, αλλά η ε, αύξηση των spreads των κρατικών ομολόγων σίγουρα επηρεάζει το τραπεζικό τομέα. Όχι μόνο, όπως λένε, πολλοί, όπως λένε πολλοί, λόγω της ε, επίπτωσης στα κρατικά ομόλογα που ε, δεν πολλούνται, αλλά και η χρηματοδότηση, το κόστος χρηματοδότησης, όπως είπατε, για το δημόσιο είναι πολύ σημαντικό. Οι επόπτες θα πρέπει να εστιάσουν στα σχέδια χρηματοδότησης των τραπεζών για να φροντίσουν ότι θα είναι αρκετά στιβαρές για να αντιμετωπίσουν και αρνητικά σενάρια ε, με τα κρατικά ομόλογα. Ευχαριστώ. Ο Σβέν Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω από την ομάδα μας ότι παρά κάποιες ε, ατυχείς δημόσιες συζητήσεις από τη δική μας προπτική τα προσόντα σας για αυτή τη θέση δεν ε, ε, είναι αμφισβητήσιμα όπως δεν υπήρχε αμφισβήτηση για μας, δεν υπήρχε αμφιβολία όσον αφορά τα προσόντα του δεύτερου υποψηφίου. Το δεύτερο είναι ότι εγώ όσο έχω εργαστεί μαζί σας, ανέκαθεν εργαστήκατε για το ευρωπαϊκό συμφέρον και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη καμία εθνικότητα. Ε, αυτό για να διορθώσω διάφορα που έχουν ακουστεί. Και σίγουρα είναι αυτά ε, δεν επηρεάζουν τη σημερινή ακρόαση. Τώρα για τη σας, το μελλοντικό σας ρόλο να δούμε κατά πόσο μπορείτε να δεσμευτείτε να εφαρμόσετε πλήρως τις ε, οδηγίες ε, περί ξεπλήματος χρήματος για τις μεγαλύτερες τράπεζες αλλά και για τις μικρότερες τράπεζες όπου ε, εσείς έχετε την ευθύνη να εξασφαλίσετε ένα ισότιμο πεδίο στην ενιαία αγορά. Στο δεύτερο, στο ρόλο σας ε, ως ε, πρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Εποπτικής Τραπεζικής Αρχής είχατε δύο ρόλους να παίξετε. Το ένα ήταν για τον τραπεζικό ρόλο και για το δεύτερο για την ΕΚΤ θα εργαστείτε δημοσιεύοντας επίσης τα αποτελέσματα των εσωτερικών δοκιμών αντοχής της ΕΚΤ, ώστε όλες οι τράπεζες του SSM να έχουν ε, στοιχεία ε, δημοσιευμένα ε, για, τους, για τα stress test, σύμφωνα με κοινούς κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την καθοδήγηση για τα... το ξέπλυμα χρήματος, από την πλευρά της Τραπεζικής Αρχής εμείς συνεργαστήκαμε για την ανάπτυξη αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, το στηρίξαμε ε, και ενώπιον της Επιτροπής σας και βεβαίως είμαι απόλυτα προσιλωμένο στο να υπάρξει επιχειρησιακή εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών και όπως είπα ήδη θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε ε, ε, κάθε ευκαιρία για να ξεκαθαρίσουμε τα ισοζύγια των τραπεζών. Και αυτό το λέω ανέκαθεν. Αυτό είναι αλήθεια για όλες τις τράπεζες. Ε, ε, το σύστημα θα πρέπει να καθαρίσει. Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και οι επόπτες να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για να τις πιέσουν ε, τόσο τις μεγάλες όσο και τις μικρότερες τράπεζες να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να μας τυπήσει επόμενη κρίση χωρίς να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε ξεκαθαρίσει τα ισοζύγια των τραπεζών από την προηγούμενη. Ναι, ρώτησα και για τις μικρότερες τράπεζες. Ναι, για μένα είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε διαφορετικές ταχύτητες προσαρμογής στις κατευθυντήριες γραμμές ε, λέει ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί η ταχύτητα ε, ανάλογα με την ε, θέση και την κερδοφορία της κάθε τράπεζας και σίγουρα θα έπρεπε να προσθέσουμε και προγράμματα για όλες τις τράπεζες ώστε να καθαρίσουν από τα μη εξυπηρετούμενα. Και τώρα, για τη δημοσίευση των stress test, των, των πορισμάτων των stress test, εδώ θα πρέπει να είμαι προσεκτικός. Γνωρίζετε ότι είμαι υπέρ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 της ε, διεμποσίευσης των πορισμάτων των stress test. Ξέρω πως αυτή η γνώμη δεν ε, βρίσκει σύμφωνη ολόκληρη την, όλους μου μάλλον τους συναδέλφους και συχνά έχω συναντήσει αντιρρήσεις και στο ίδιο το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Όμως, ε, όπως σας είπα, για μένα είναι απαραίτητο να έχουμε το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας. Ευχαριστώ κύριος Παπαδημούλης. Κύριε Ενρία, να σας καλωσορίσω και στην Επιτροπή μας. Είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω την παρουσίαση που μας κάνατε στην ε, συνεδρία των συντονιστών in camera και θέλω να πω ότι η εντύπωση που μου προκάλεσε η παρουσίασή σας ήταν εξαιρετικά θετική δείξατε έναν υψηλό επαγγελματισμό και μια αίσθηση υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Και νομίζω ότι ορισμένα σχόλια που δυστυχώς είδα στον τύπο που επηρεάζουν και προβλέπουν το πόσο καλά θα κάνετε τη δουλειά σας από το σε ποιο κράτος μέλος ανήκετε και από ποιο κράτος μέλος προέρχεστε, νομίζω ότι δεν υπηρετούν ούτε την ε, αξιοπιστία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, ούτε την ευρωπαϊκή ιδέα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τρία πράγματα, επειδή έχετε και την εμπειρία, καθώς ήσασταν πρόσφατα ένας ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Το πρώτο πράγμα, πριν από εσά ήταν εδώ η κυρία Νουή και πιθανότατα θα τη διαδεχτείτε εφόσον το Ευρωκοινοβούλιο, και σας το εύχομαι, ψηφίσει θετικά για την υποψηφιότητά σας. Μας είπε ότι είσαστε ως θεσμός και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο SSM θερμοί υποστηρικτές της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ενοποίησης και με το ίντις, καθώς έχει μειωθεί σημαντικά το ρίσκο και είναι ώρα να μοιραστεί να αμοιβεοποιηθεί και το, το ρίσκο. Θα ήθελα τη δική σας γνώμη. Γνωρίζω ότι είναι πολιτική απόφαση, αλλά αν εσείς οι ειδικοί ορθώσετε περισσότερο ε, τη δική σας φωνή, αυτή η ατελής τραπεζική ενοποίηση ίσως προχωρήσει ταχύτερα και προλάβουμε ζημιές από την επόμενη κρίση, καθώς οι κρίσεις κάνουν κύκλους. Το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω, εκτός από την ατελή τραπεζική ενοποίηση και την ανάγκη να καλυφθούν ελλείμματα, είναι το ατελές σύστημα ελέγχων. Πώς πέρασε κάτω από το ραντάρ όλων αυτών των θεσμών των ελέγχων το σκάνδαλο Κούμεξ ή προηγούμενα σκάνδαλα που είχαν άλλα ονόματα. Panama Papers, Paradise Papers, πώς μερικές δεκάδες whistleblowers, δημοσιογράφοι, βρίσκουν πράγματα που δεν μπορούν να βρουν ισχυρές λεγκτικές αρχές. Και το τρίτο, επειδή έχετε επανειλημμένα μιλήσει για την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας, θα ήθελα να μου πείτε από το πόστο του επικεφαλής του SSM, εφόσον το αναλάβετε, τι σκοπεύετε να προτείνετε και να κάνετε για να ενισχυθεί η διαφάνεια, καθώς οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια και έχουν μεγάλη δυσπιστία. Thank you very much. Let me start. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω με το θέμα της ε, τραπεζικής ε, ολοκλήρωσης. Ε, εκφράστηκα πολλές φορές υπέρ αυτού του σχεδίου και για πολλούς ε, λόγους σε πολιτικό επίπεδο συζητάτε πάρα πολύ το θέμα της ενοποίησης ε, του ρίσκου και της προστασίας των καταθέσεων, αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε στο αυτού μας ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες ε, που θα υπαχτούν σε καθεστώς ε, εξυγίνησης θα πρέπει να τηρήσουν αυτούς τους όρους που έχουν στόχο να επιβάλλουν κάποιες ε, υποχρεώσεις στις τράπεζες. Το πρόγραμμα προστασίας των καταθέσεων πρέπει ε, να προσφέρει επαρκείς εγγύησεις ε, στους καταθέτες. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές ε, επιπτώσεις ε, του σχεδίου ε, έντις και είναι μικρό το κόστος. Μιλήσατε για τη τραπεζική ολοκλήρωση. Σήμερα όλες οι, όλες οι προστατευτικές δράσεις που εφαρμόστηκαν μετά την κρίση έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν ε, τις συνέπειες ε, των ε, κρίσεων. Και αυτό θα επέτρεπε και τον επιμερισμό του κινδύνου. Κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν είμαι υπέρ του σχεδίου Καταλαβαίνω ότι γίνεται μια συζήτηση για την, το καταπαρισμό και τη μείωση των κινδύνων. Ε, πάντα εργαστήκαμε με οδικούς χάρτες και αυτό μας ε, επέτρεψε να ε, ε, επιτύχουμε και τους δύο στόχους σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι ε, μετά την κρίση και τις καταστροφικές συνέπειες βλέπουμε ακόμα ε, τράπεζες ε, και τη φήμη τους να διακυβεύονται με αυτά τα σκάνδαλα. Για μένα το σημαντικό για τις εποπτικές αρχές είναι η εσωτερική διακυβέρνηση, η διαχείριση του κινδύνου. Αυτή είναι η τομής στους οποίους οι επόπτες μπορούν πραγματικά να προσφέρουν προστιθέμενη αξία προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των αξιών στα πλαίσια του τραπεζικού συστήματος. Πρέπει να εργαστούμε στεναρά και αυτή είναι η δέσμευσή μας. Ε, αν εγκριθεί η υποψηφιότητά μου, πρέπει και στο SSM και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα να εργαστούμε προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι, δύο στόχοι και με την χρησιμοποίηση προληπτικών εργαλείων ε, σε διάφορα ε, επίπεδα. Αναφέρεται επίσης το θέμα της διαφάνειας καταλαβαίνω προς το SSM, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν δεσμευτεί ε, υπέρ της διαφάνειας στα πλαίσια της διεξαγωγής ε, του, των εργασιών τους ε, και συμφωνώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε το ανώτατο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και εγώ θα ε, φροντίσω να δεσμευτώ για την επίτευξη ε, αυτών των στόχων στα πλαίσια των νέων μου καθηκόντων αν διοριστώ. Ε, ανέφερα ήδη το θέμα του δεύτερου πυλώνα που παίζει πρωταρχικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη σχέση των επενδυτών και των τραπεζών. Ευχαριστώ πολύ. Η Ντανούτα Χούμπνερ. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν κοινό νόμισμα. Πρέπει να μπουν στην Τραπεζική Ένωση, να τους ενθαρρύνουμε ή όχι. Θα θυμάστε ότι το 2014 νομίζω η Κεντρική Τράπεζα της Δανίας ενθάρρυνε την κυβέρνηση να προσχωρήσει θεωρώντας ότι θα ωφελούσε τη Δανία αλλά πριν από λίγο καιρό η κυβέρνηση ε, το ανέβαλε για το 2019 μετά τις εκλογές. Τώρα το σκάνδαλο της Ντάνσκα ε, επανεκκίνησε τη συζήτηση και η δανεική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προσχωρήσει. Και η επιστολή της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και στην ΕΚ το καλοκαίρι, οι ε, Υπουργοί Οικονομικών τον Ιούλιο Ε, είδαν την πρόθεση προσχώρησης. Η συμμετοχή στην Τραπεζική Ένωση θα μπορούσε τώρα να λύσει κάποια προβλήματα του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα την καταπολέμηση του ξεπλήματος, βελτίωση της εποπτείας, αντιμετώπιση της διαφθοράς ε, στον τραπεζικό τομέα, τα σκάνδαλα. Ε, τι λέτε, η προσχώρηση στην ε, Τραπεζική Ένωση θα ήταν καλή ή θα ήταν περισσότερη δουλειά για σας, θα έδινε κάποια ωφέλη, υπάρχει προστιθέμενη αξία αν αυτές οι χώρες μπουν στην Τραπεζική Ένωση πριν μπουν στην Ευρωζώνη. Θα ήταν καλό κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Καταρχήν η απόφαση συμμετοχής στην Τραπεζική Ένωση είναι απόφαση των κρατών μελών που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Εκείνοι θα επιλέξουν αυτή τη μορφή ε, ε, της εισόδου. Είναι η δική τους απόφαση. Από την πείρα μου στην τραπεζική αρχή συχνά ε, ασχολήθηκα με διαμεσολαβητικές διαδικασίες μεταξύ ε, ιδρυμάτων που ήταν χωρών στην Τραπεζική Ένωση και άλλων. Η αντίληψή μου είναι ότι ε, μάλλον, αν διοριστώ στη θέση δεσμεύομαι να φροντίσω ότι θα σέβομαι την απαραίτητη ισορροπία που θα επιτρέπει κοινέ αποφάσεις και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και στις τράπεζες για τις οποίες έχει ευθύνη ο SSM. Αλλά είναι άλλη υπόθεση αν κάθεται κανείς στο τραπέζι και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για τις τράπεζες που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στις τοπικές, και εσωτερικές αγορές. Υπάρχει λοιπόν προστιθέμενη αξία που με ρωτάτε και αν προκειμένου περί της Βουλγαρίας ε, ε, ε, διατυπωθεί αίτημα, ο SSM και η ΕΚΤ e θα κάνουν το καλύτερο για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και να εξομαλυνθεί η προσχώρηση στην Τραπεζική Ένωση της Βουλγαρίας. Ευχαριστώ, Γιάκοπ Φον Βάιτσέκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ανρία, ένα-δύο σύντομες ερωτήσεις μόνο. Πρώτη είναι, πιστεύετε πως το ενιαίο σημείο ε, στρατηγικής εξυγίανσης που έχουν οι περισσότερες μεγάλες τράπεζες ε, μετά το Brexit και με το κάπως ε, πιο τεταμένες υπερατλαντικές σχέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Δεύτερη ερώτηση είναι κατά πόσο θεωρείτε πως η εποπτική διακριτική ευχαίρεια θα πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο ώστε να βοηθηθούν οι πιο δύναμες τράπεζες να οικοδομήσουν αρκετά αντικυκλικά, αντικυκλικούς φραγμούς συμπεριλαμβανομένων των stress test. Και έπειτα υπάρχει λόγος για να εφαρμοστεί η τεχνολογία RedTech από, περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Το, το ενιαίο σημείο εισόδου είναι ακριβώς ένα πρότυπο που απαιτεί πολύ συντονισμό εξάντε όσον αφορά την προετοιμασία και εξπόστο όσον αφορά την ε, λειτουργία του συστήματος εξυγίανσης ώστε να είναι αυτό αξιόπιστο. Σε πολλές περιπτώσεις ε, η ε, Αυτό συνδέεται και με τον, ε, το σύστημα της ε, εγγύησης του, της, της τράπεζας, αυτό εξαρτάται από το πώς ε, θα εξελιχθεί η κίνηση, δηλαδή ανάντι, κατάντι ε, και ούτω καθεξής. Νομίζω πως το Brexit και οι υπερατλαντικές τεταμένες σχέσεις που αναφέρατε δεν είναι το κύριο πρόβλημα εδώ, γιατί σε κάποιο βαθμό όπως ε, θα γίνει θα είναι πλέον τρίτη χώρα σε λίγους μήνες και βέβαια η ΕΠΑ είναι ήδη τρίτη χώρα. Άρα Εάν γίνουν δεκτές οι, τράπεζες, οι προτάσεις της ε, IBU και γίνουν δεκτές οι προτάσεις που κάνει ήδη στην τράπεζα, έχουμε ε, ε, έναν μηχανισμό που θα μπορέσει να φέρει την εξυγίανση εντός της εγχώριας δικαιοδοσίας. Οπότε η έκδοση SP δεν είναι τόσο σημαντική. Όσον αφορά την διακριτική εποπτική ευχέρεια, να σας πω ειλικρινά ότι αν εσάς αναφέρεστε στους αντικυκλικούς φραγμούς, αυτοί θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από την ε, μικροπροληπτική ε, ε, πρόβλεψη θα έπρεπε να είναι κάτι περισσότερο, αλλά έχετε δίκιο πως κάποιες φορές οι μικρές τράπεζες θα πρέπει να εξετάζονται πιο προσεκτικά, διότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα δραστήριες σε πολύ κυκλικές αγορές, όπως ας πούμε η αγορά ενυπόθηκων δανείων που είναι σημαντική. Η εφαρμογή λοιπόν αυτών των φραγμών για μικρές τράπεζες μπορεί να χρειαστεί να γίνει σύμφωνα με την διακριτική ευχέρεια. Να δω ότι δεν βγάζω τα γράμματά μου. Α, ναι, το RegTech. Είπατε πως ε, είναι μια ενδιαφέρουσα, ένα ενδιαφέρον εργαλείο Εγώ θα πρότεινα να διερευνηθεί, να διερευνηθεί το κατά πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο. Στην ε, EBA έχουμε, διερευνήσει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με τις, τα αιτήματα των ε, νεοϊορκέζων ε, συνεργατών μας. Είναι πολύ δύσκολη όμως η επαλήθευση και αυτό ε, θα μπορούσε κάπως να ελαφρύνει τη διαδικασία. Αυτή η, διαδικασία, αυτό το εργαλείο, το RegTech, θα μπορούσε να διευκολύνει ε, την όλη διαδικασία, θα μπορούσε να είναι μια σημαντική εξέλιξη και θα πρέπει να διερευνήσουμε το ε, τομείς για περαιτέρω χρήση του εργαλείου αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. τελειώσαμε νομίζω ακριβώς την ώρα. Βεβαίως υπάρχει catch the eye, εάν κάποιος θέλει το λόγο. Διαφορετικά, να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση και τώρα να ε, ολοκληρώσουμε αυτή την ακρόαση και να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.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

Dear colleagues, let's start. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, να ξεκινήσουμε με μία δοκιμή παρακαλώ. Για ψηφίστε. ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα. Μπορούμε να κλείσουμε τη δοκιμή μας και η πρώτη ε, ψηφοφορία είναι η έγκριση του διορισμού στην Προεδρία του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μόλις ακάναμε την ακρόαση, είναι μυστική ψηφοφορία, μπορείτε να ψηφίσετε. Vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. 42 υπέρ, μία κατά, 9 αποχές. Συγχαριστήρια στον Ανδρέα Ενρία. Δεύτερη ψηφοφορία αφορά το σχέδιο έκθεσης του Μπέτ Λούκε για τα καλυμμένα ομόλογα. Ξεκινάμε με την οδηγία. Σωστά. Ωραία. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική σ με προφορική τροπολογία της ομάδας των σοσιαλιστών. Πρώτα η ε, προφορική υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D. Α, συγγνώμη, έχετε το λόγο. Η κυρία Μπερές. Συγγνώμη, αλλά εγώ θεωρώ πως εφόσον δεν πέρασε η προφορική τροπολογία, υπάρχουν τρεις τροπολογίες που δεν καλύπτονται από τη συμβιβαστική δηλαδή οι 126, 175 και οι 178. Μπορείτε να μου πείτε πάλι τα αριθμού των τροπολογιών. 146. Μάλιστα. 175. Ναι, αυτοί συμπεριλαμβάνονται στην συμβιβαστική F. Εδώ είναι η 146 που θα έπρεπε να ψηφιστεί. Μάλιστα, ζητάτε χωριστή ψηφοφορία για την 146 οι σοσιαλιστές. Ο εισηγητής παρακαλώ, όχι, ε, είμαι κατά αυτής της άποψης. Η τροπολογία των σοσιαλιστών εξετάστηκε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των σκιωδών, δεν ε, υπερψηφίστηκε και βασικά ε, καλύφθηκε από τη συμβιβαστική και οι ομάδες συμφώνησαν να μην συμπεριληφθεί στη συμβιβαστική, άρα καλύπτεται. Ο κύριος Σάντ, παρακαλώ. Sorry. Um, στη διάρκεια της συνεδρίασης των σκιωδών ήταν σαφές ότι χρειαζόταν ψηφοφορία από αυτής εδώ. Ε, χρειαζόταν ψηφοφορία διότι η συμβιβαστική δεν, το, δεν την κάλυπτε θέλαμε λοιπόν να ψηφιστεί χωριστά. Thank you. Sorry, honestly, it's not the... Κοιτάξτε, ειλικρινά δεν είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα ζητά χωριστή ψηφοφορία που καλύπτεται από μια συμβιβαστική. Δεν είναι και το τέλο του κόσμου που ψιάζουμε πω θα είναι και η ίδια πλειοψηφία. Δεν είναι και τόσο σπουδαίο, οπότε α το ψηφίσουμε χωριστά. 146 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και πάμε στη συμβιβαστική D υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ή e, υπέρ, κατά, ε, ε, ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική F με προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Ψηφίζουμε πρώτα για την προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται. Ψηφίζουμε στη συμβιβαστική χωρίς την προφορική. Η κυρία Μπερές. Ναι, θα ψηφίσουμε την 175 και την 178 χωριστά. Θέλετε, μάλιστα. Ναι, συμβιβαστική F χωρίς την προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψηφίστε παρακαλώ. Vote is Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 26 έναντι 24 και τώρα ψηφίζουμε την 175 χωριστά 175 υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται Τέλος. Απορρίπτεται. 178 είπατε οι άλλοι, υπέρ, κατά, απορρίπτεται νομίζω, εκτός αν θέλετε και εδώ έλεγχο ηλεκτρονικό, όχι. Ωραία λοιπόν, πάμε στη συμβιβαστική G, υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 259 υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται. Vote is Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική K. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική L με προφορική. Πρώτα ψηφίζουμε την προφορική. Υπέρ. Κατά. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 25 προς, 100 προς 22 υπέρ. Τώρα L. Η συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ο μικρόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 34 υπέρ, 16 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγήτη. Α, όχι, πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων επί τη βάση της έκθεσης όπως υιοθετήθηκε στην Επιτροπή. Νομαστική κλίση άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται υπάρχει ειδική πλειοψηφία. Οπότε τώρα περνάμε συγχαρητήρια, περνάμε στον κανονισμό και ψηφίζουμε πρώτα την τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, έχω λάθος κατάλογο ψηφοφορίας. Just a second. Okay, yes. Um, Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά Έλεγχος για τη 15 άρχεται. Τέλος. Απορρίπτεται 22 προς 20. Αν μπλοκ ψηφίζουμε τις 38 και 39. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 16. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται τέλος ψηφοφορίας ε, ε, εγκρίνεται 26 ψήφοι υπέρ 24 κατά τροπολογία 17 υπέρ κατά το ΕΛΚ υπέρ μάλιστα αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά α, έλεγχος ηλεκτρονικός άρχεται τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται η τρία έχει αποσυρθεί. Η τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονικός για τη 19 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για την πρόταση της Οικομισιόν όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική κλίση άρχεται. πέρας. 45 υπέρ, 5 κατά μία αποχή. Ψηφίζουμε για την έναρξη διαπραγματεύσεων επί τη βάση της έκθεσης όπως υιοθετήθηκε στην Επιτροπή με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. 44 υπέρ, 6 κατά. Και τώρα να συγχαρώ τον εισηγητή Ε, σχέδιο έκθεση της Μπάρμπαρα Κάμπελ για την ετήσια έκθεση τη Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ξεκινάμε με την τροπολογία 20. Okay, sorry. Amendment 20. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία επί της 21 πέρας απερίφθη 22 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία επί της 22 Πέρας. Ε, ισοψηφία απορρίπτεται 24 από 24. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ε, ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 28 υπέρ 17 κατά πάμε στη συμβαστική Β όπου πρέπει να πω ότι ο εισηγητής ενημέρωσε τη γραμματεία ότι το Α, α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Όχι, ψηφίζουμε την τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 29 υπέρ, κατά, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία επί της 29. Πέρας. Απερίφθη. Τώρα, συμβιβαστική Β. Έλεγα ότι ε, ενημερώθηκε η γραμματεία από τον εισηγητή ότι το περιεχόμενο της, ε, κατά λάθο μπήκε μια τροπολογία στη συμβαστική Β. Έπρεπε να καλύψουμε την 13 ε, ίντα χωρίς τη διατύπωση της τελευταίας παραγράφου. Το τελευταίο της 13 ΙΝΠΑ δεν έχει συμπεριληφθεί στη συμβιβαστική τροπολογία. Γι' αυτό το κείμενο που αρχίζει καλή την EIB λαμβάνοντα υπόψη και λοιπά μέχρι συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, αυτό διαγράφεται. Αυτή είναι η ανακοίνωση του εισηγητή. Με αυτή τη διευκρίνηση λοιπόν ψηφίζουμε τη συμβαστική Β υπέρ κατά έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία τη συμβαστικής Β. Πέρας. Δεκτή. 30 προς 19. Πάμε στην τροπολογία 37. Όχι, 35. Όχι, βλέπω ότι έχει ε, αποσυρθεί. Είχα δίκιο λοιπόν, έχει αποσυρθεί. 37. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 έχει αποσυρθεί και αυτή, οπότε πάμε στο αρχικό κείμενο. Της παραγράφου 4 υπέρ. Κατά. Έλεγχος στο αρχικό κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Τροπολογίες 39 και είναι τα ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Παράγραφος 7 τα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αυτά καλύπτονται. Πάμε στη 45. Θέλετε να γίνει έλεγχος ε, ηλεκτρονικός στη 43. 43. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλμαρ, καλώς ήρθες στην ΕΚΟΝ. Πέρας. Δεκτή. 28 προς 23. Πάμε τώρα στη 45. Υπέρ. Κατά αποχές Νομίζω η ίδια πλειοψηφία, αλλά ήταν πολύ κοντά. Ψηφίζουμε τη 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω να δούμε τη 49 ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Την 50 ψηφίζουμε. Πέρας δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή αρχικό κείμενο ε, υποτομέας ε, δεκτό 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό 60 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία επί της 60 νέος συνδυασμός είναι αυτός πολιτικών ομάδων πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται 26 προς 21 υπέρ. Ε, συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στο budget 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Budget παράγραφος 16, budget 16. Budget παράγραφος 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 66 υπέρ έλεγχος στην 66, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 72 υπέρ ε, κατά απορρίπτεται όλε σαν μπλοκ. <laughs> Σα αρέσουν οι τροπολογίε. 73 ε, απορρίπτεται, 76 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται, 78 υπέρ κατά ε, απορρίπτεται, 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο ε, Τέσσερα υποπαράγραφος ε, υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας δεκτό 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο παράγραφος 8 υπέρ κατά αποχές δεν είδα τα χέρια πολλών ομάδων. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία από το αρχικού κειμένου του παραγράφου 8. Πέρας. Δεκτό. Να φαίνονται τα χέρια. Τροπολογία 85. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο στο υποτομέα 5 υπέρ κατά αποχές δεκτό 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο παράγραφος 9 υπέρ κατά αποχές δεκτό 89 υπέρ κατά αποχές δεκτή 91 υπέρ κατά έλεγχος της 91 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 26 προς 24. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Παράγραφος 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 93 υπέρ. Κατά Άρχεται η ψηφοφορία επί της 93. Πέρας. Ε, ισοψηφία. Απορρίπτεται λοιπόν. 94 υπέρ κατά έλεγχος στην 94. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 29 προς 22. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή. Budget παράγραφος 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 19 υπέρ. Κατά έλεγχος. Budget 19 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 102 υπέρ κατά αποχές δεκτή 103 υπέρ κατά έλεγχος στην 103 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο ε, στο 6 υποτομέα ε, υπέρ κατά 107 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπό παράγραφος 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά έλεγχο στην 110 άρχεται η ψηφοφορία 110 πέρας δεκτή 24 προς 19, 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 112 υπέρ κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ελέγχουμε 112, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 12 υπέρ. Κατά να φαίνονται τα χέρια, αλλά το ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα. Οι σοσιαλιστές είναι ε, κατά. Πέρας. Δεκτό. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 132 υπέρ κατά έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία 25-25 απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Ή. E, υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα παράγραφος 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή παράγραφος 5 υπέρ κατά έλεγχος είναι τα παράγραφος 5 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απερίφθη με μία ψήφο διαφορά 24 προς 23 είναι τα 8 υπέρ έλεγχος ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέρας δεκτή η 30 προς 19 είναι τα 11 υπέρ κατά έλεγχος Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι τα 11. Πέρας. Ισοψηφία 26-26. Απορρίπτεται. Budget, παράγραφος 15. Περίεργα πράγματα. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Budget 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές δεκτή. Budget 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, budget 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή, 158 υπέρ κατά αποχές έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία επί της 158. Πέρας. Απερίφθη 23 προς 28. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο παράγραφος 17 υπέρ κατά αποχές δεκτό budget παράγραφος 10 υπέρ κατά αποχές δεκτό budget 11 υπέρ κατά αποχές δεκτό τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο αιτιολογική α υπέρ κατά αποχές δεκτό 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή μπει αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό τροπολογία 7 υπέρ κατά έλεγχο στην 7 άρχεται η ψηφοφορία και συγχαρητήρια στον καταθέσαντα αυτή την τροπολογία που έγινε Βέλγος Υπουργός Άμυνας. Τέλος της ψηφοφορίας. Νιώθω πιο ασφαλής τώρα. Πέρας λοιπόν. Απερίφθη. Πάμε τώρα στο αρχικό κείμενο, παράγραφος B, όχι, όχι, για έκανα την 8 πρέπει να ψηφίσουμε, όχι την 8. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 9 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 10 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 11 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Είπαμε τι ισχυρός που είναι, όλες περνάνε, περνάνε, ασκούνται πυροές. 12 ε, υπέρ, κατά έλεγχος στην 12 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απερίφθη αρχικό κείμενο αιτιολογική υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτό ε, ε, ε λογική D υπέρ κατά αποχές δεκτό το αρχικό κείμενο ε, αιτιολογική ε υπέρ κατά αποχές δεκτό 13 υπέρ κατά έλεγχο στη 13 άρχεται η ψηφοφορία η 13 πέρας απορρίφθηκε 28 προς 24 υπέρ. 14, τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ε, τώρα πάμε σε αναφορικές ε, προτάσεις. Ε, θέλετε να πάμε από το 1 στο 9 μπλοκ. Ναι, όλες μαζί, από το 1 μέχρι το 9. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά αρχικό κείμενο ε, το 10 κατά αποχές έλεγχος έλεγχος πέρας δεκτό ε, τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ονομαστική κλίση επί του κειμένου όπως ετροποποιήθη άρχεται η ψηφοφορία The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 9 κατά 9 αποχές, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πάμε τώρα στη Βάνα Μαλέτιτς για τις κοινέ διατάξεις, τον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις. Αρχίζουμε με την τροπολογία 20. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές έλεγχος την 23 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας απορρίπτεται 28 με 23 ε, τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά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 εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος δεν είδα καλά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 27 προς 23. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40. Και 41. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρες; Απορρίπτεται. 29 προς 22. 42. Τρει ήταν οι τροπολογίε. Άρα περνάμε στην 7. Ε, Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Έλέγχο για τη 43. Άρχεται η ψηφορία. Πέρες. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για τη 44 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρες. Απορρίπτεται. 45. 45 και 46 είναι ίδιες. Υπέρ. Κατά. Απο... Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 προς 23, με 23, ε, ε, τροπολογία 8, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 47, υπέρ κατά Α, η 47 καταπίπτει. 48 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφορία. Πέρες. Απορρίπτεται. 28 προς 23. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 50. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 27 προς 24. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν λοιπόν στη 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 προς 24. Ε, Τροπολόγια 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28, 58 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκτός αν θέλετε έλεγχο, έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήταν η 11, περνάμε στην 61, υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 61. Πέρες. Απορρίπτεται. 26 προς 24. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με, ε, οριακά. Με την ίδια ε, ψηφία με προηγουμένως. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 63 απορρίπτεται. Ναι, άρα πρέπει να περάσουμε στην 64. Να κάνουμε έναν έλεγχο για την 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 22, προς 22. Περνάμε στην 66 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 66 Περβάνσε για την τροπολογία σου πρόκειται πέρας απορρίπτεται 28 προς 22 ε, αποσύρεται αποσύρεται περνάμε στην 61 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω το ECR. Τι αποφασίζει. Κατά. Άρα απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 85 υπέρ. Το ΕΛΚ είναι υπέρ ή κατά. Κατά. Έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται.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 αποχές απορρίπτεται, 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 109 109 υπέρ κατά ναι, καταπίπτει η 109, σωστά. 110 υπέρ κατά έλεγχος για την 110 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 και 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά άλλη είναι υπέρ ή κατά. Απορρίπτεται 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 28 προς 20, 127. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 125 και 126 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 και 129 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 132 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 133 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 134 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 135, 136 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 137 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 138 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 139 υπέρ, κατά αποχές η Άλντε είναι κατά τη 199. Ε, απορρίπτεται. 1. Υπέρ κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για τη 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 προς 24. 3. Υπέρ. Κατά. Γιάλντε. Κατά. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 12 και 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά Έλεγχος γιατί τη 4, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ε, ψήφο διαφορά 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παρατήματα 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφορία για το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 28 υπέρ, 24 κατά, 0 αποχές, εγκρίνεται, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έχουμε και ένα δεύτερο μέρος. Δεύτερη έκθεση της ε, κυρίας Μαλέτιτς για τη συζήτηση για την κατάσταση της Ευρώπης. Συμβαστική Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β με μια προφορική ε, τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Δ υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ε υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 40 υπέρ, 7 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια ε, στην εισηγήτρια. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο. Με ε, ε, νέα με 1 και η τακτική συνεδρίαση της ΕΚΟΝ τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε στις 9 ακριβώς, να είστε στην ώρα σας. Μα πάντα ξεκινάμε στην ώρα μας. Διαφορετικά θα υπάρχει επικάλυψη με την επόμενη συνεδρίαση. Πρέπει να ξεκινήσουμε στην ώρα μας. Ε, Δευτέρα ε, στις 3 και την Τρίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, λίγη συνεδρίαση.